Hello, everyone. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάει η συνεδρίαση. Σε ό,τι αφορά την Μέσια Διάταξη, δυστυχώς ε, χρειάστηκε να ακυρώσει την ε, συμμετοχή του συνεδρίασή μας ο Αντιπρόεδρος Επιτροπής, ο κ. λόγω προβλήματος υγείας, δυστυχώς. Τελευταία στιγμή, λοιπόν, ακυρώθηκε η παρουσίαση παρουσία του εδώ σήμερα και χρειάστηκε να αλλάξουμε την μερίσια διάταξη. Θα μπορέσουμε να συζητήσουμε κάποιες αντιρρήσεις. Ε, δουλειά έχουμε να κάνουμε τόσο ή άλλως, δεν σημαίνει ότι θα ε, ελαφρυνθεί πολύ η μερίσια διάταξη. Λοιπόν, βγάζοντας έξω την παρουσία του κ. Σεύκοβιτς, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη κατά τα υπόλοιπα σημεία. Αν έχετε στο φάκελό σας ε, την έκθεση από την αποστολή τη ΕΝΒΗ σε Ταλίν και Βόρεια στον 22-24 Μάιο. Γιατί άργησε, δεν ξέρω. Τέλο πάντων θα το δούμε αυτό. Ε, έχουμε 21 γλώσσες διερμηνία σήμερα και ως συνήθω. Ηλεκτρονικό θα λάβετε το φάκελο της συνεδρίασης. Ε, σε ό,τι αφορά τις ε, ανακοινώσεις για τους ε, συντονιστές, αν δεν έχω κάποια αντίρρηση, θα θεωρήσουμε ότι οι συστάσεις τους εγκρίνονται. Επόμενη αναφορά μας στις διοργανικές διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε δύο-τρία πραγματάκια. Πρώτον, μηχανισμός ε, παρακολούθησης και αναφοράς για τις εκπομπές αέριων θερμοκηπίου. Ελήφθησαν υπόψη ε, τα συμπέρασματα των τεχνικών συναντήσεων, ιδίων ε, σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση και την ευελιξία. Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για αυτά τα σημεία, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμη συμφωνία Κοινοβούλιο και Συμβούλιο διαφωνούν μεν για κάποια κρίσιμα σημεία, αλλά οι συζητήσει ήταν επικοδομητικέ. Αυτή είναι η δική μα άποψη ω Κοινοβούλιο στο δεύτερο του διάλογο για το effort sharing. Θα εξεταστούν άλλα τεχνικά ζητήματα στην επόμενη συνάντηση τεχνικού επέδου πριν τον τρίτο τριμερή διάλογο. Για το Λούλου Σιεύκουν το επόμενο θέμα. Είχαμε το δεύτερο άτυπο τριμερή διάλογο στις 22 Νοεμβρίου. Κοινοβούλιο και Συμβούλιο συμφώνησαν σε ορισμένα ζητήματα τα οποία είχαν ήδη εγκριθεί σε τεχνικό επίπεδο και σε κάποια άλλα θέματα επίσης. Για τα πιο λεπτά από πολιτικής πλευρά ζητήματα όπως είναι η δυνητική ευελιξία για τη δασική γη και το θέμα της διακυβέρνησης για την αναθεώρηση κάποιων επιπέδων αναφοράς για τα δάση Έγινε συζήτηση για αυτά τα θέματα και οι διαπραγματευτές θα αφήσουν την περαιτέρω εξέταση των θεμάτων σε τεχνικό επίπεδο πριν την τρίτη συνεδρίαση του μέρους διαλόγου για τις 14 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο έχει προβλεφθεί αυτή. Um, σε ό,τι αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες στον τομέα της ε, υποβολής περιβαλλοντικών αναφορών, πρώτος και τελευταίος του Μέρου διάλογος για την απόφαση σε ό,τι αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες στις 22 Νοεμβρίου και αυτός, το μέρης διάλογος, οι δύο συνομοθέτες είχαν ε, σχεδόν την ίδια άποψη επί των τροπολογιών, επομένως εύκολα κατέληξαν σε μια προσωρινή συμφωνία. Η δική προσοχή δόθηκε στην έναρξη ισχύω της απόφασης. Διότι υπάρχουν κάποια άτομα που θα πρέπει να συσχετιστούν με τις διατάξεις των διοργανικών διαπραγματεύσεων που αφορούν το ETS. Λύθηκε το ζήτημα με τη διασύνδεση της απόφασης με το ETS, όμως αποφασίστηκε αναβολή της ε, ψηφοφορίας μέχρι να υπάρξει συμφωνία για τα θέματα του, πακέτου για τα απόβλητα, ώστε να υπάρχει νομική συνέπεια. Που σημαίνει ότι εμείς στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε κατά πάσα πιθανότητα τον Ιανουάριο. Και τώρα περνάμε στο σημείο 5. Ευρωπαϊκή στρατηγική για ΕΦΗ συστήματα μεταφορών, συνεργατικά. Έχουμε την εισηγήτρια εδώ, την κυρία Σάλντε Μόζε. Είναι έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας Επιτροπής Μεταφορών. Δεν καθυστερώ άλλο εγώ. Δίνω το λόγο αμέσω στην εισηγήτρια και σε όποιον άλλο θέλει το λόγο. Πρώτα η κυρία Σαλτεμόζε. Ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένω να βάλετε όλοι τα ακουστικά σας, γιατί σήμερα θα σας τα πω στα δανέζικα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εδώ είναι να γνωμοδοτήσουμε στην Επιτροπή Μεταφορών, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την εβδομάδα ε, γιόρτασε την πρώτη εβδομάδα της, την πρώτη χρονιά της ε, στρατηγικής ε, για χαμηλών εκπομπών μεταφορές. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο των αυτοματοποιημένων εφιών μεταφορών. Τα συνεργατικά εφή συστήματα μεταφορών όπως τα ονομάζουμε. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε εμείς εδώ είναι να βοηθήσουμε ώστε αυτή η τεχνολογία να μας δώσει νέες δυνατότητες στο πλαίσιο του τομέα των μεταφορών, να έχουμε νέες υπηρεσίες. Θα είναι ένας από τους κινητήριους μοχλούς της επανάστασης στον τομέα των μεταφορών. Θα μας επιτρέψει τεχνολογικές καινοτομίες, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, Φυσικά και η ψηφιοποίηση θα επηρεάσει και τον τομέα των μεταφορών, αλλά αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό και που πρέπει να τονίσουμε και είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό είναι το θέμα της ανάπτυξης της ε, απασχόλησης ε, και στον τομέα των μεταφορών. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη νέα τεχνολογία ώστε να μπορέσουμε να τονίσουμε την βιωσιμότητα του τομέα των μεταφορών. Αυτές οι νέες ψηφιακές δυνατότητες πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτή, αυτόν τον χαμηλών εκπομπών ε, αυτή τη χαμηλών εκπομπών κινητικότητα που όλοι την επιθυμούμε. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ σημαντικό, ε, σημαντική δυναμική μείωση των οξυδίων του αζότου, του διοξυδίου του άνθρακα, τη συγκέντρωση ε, του όζοντος και της συγχωρήπανσης. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία μπορούν να συνδυαστούν με τις ψηφιακές τεχνολογίες που θα δώσουν τη δυνατότητα στα λεωφορεία τα αυτοκίνητά μας να μπορέσουν να επικοινωνούν μεταξύ τους για να γίνεται καλύτερη διαχείριση ε, της ε, κυκλοφορίας, ε, μείωση της συγχωρήπανσης, μείωση των εκπομπών, των λεωφορείων, των αυτοκινήτων κλπ. Αυτό σημαίνει ότι αν μπορούμε καλύτερα να διαχειριστούμε όλα αυτά, θα έχουμε πολύ μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Γι' αυτό ακριβώς η Επιτροπή Περιβάλλοντος πρέπει να γνωμοδοτήσει. Αυτή η πτυχή πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είναι πολύ σημαντική αυτή η στρατηγική. Θέλουμε να αυξήσουμε τι θέσει απασχόληση. Θέλουμε να πρωτοστατεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στον καθορισμό των προτύπων για αυτά τα ευφυή e συστήματα μεταφορών. Αλλά νομίζω ότι το βασικό μας καθήκον εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο να είναι ένα ποιοτικό εργαλείο, εύχριστο, σε σχέση με την ε, προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, γιατί μειώνοντας τις εκπομπές αερίων, ε, προφανώς αυτό θα έχει μια σημαντική συνέπεια στη δημόσια υγεία, γιατί θα μειωθούν τα οξύδια του αζότου, του διοξιδίου του άνθρακα και με τη μείωση της συγχωρήπανσης, αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να υπάρξουν θετικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ενδυνάμει πλεονεκτήματα προκειμένου να συνεχιστεί η ανάπτυξη αυτών των εφιών συστημάτων. Υπάρχει και το θέμα της οδικής ασφάλειας βέβαια και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα αυτοκίνητά μας ε, δεν θα πατάνε κόσμο στο δρόμο, ήδη είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας ε, σε σχέση με τη στρατηγική αυτή που μας δίνει νέες δυνατότητες, αλλά πρέπει να είμαστε συνάμα και προσεκτικοί. Πρέπει να λέμε στη γνωμοδότησή μα ότι οι χαμηλέ εκπομπέ πρέπει να είναι ένα στόχος τον οποίο θέλουμε να εκπληρώσουμε κάθε φορά που ξεκινούμε αυτή την προσπάθεια ανάπτυξη των συστημάτων μεταφορών των εφιών δεν είναι μόνο ένα ζήτημα ανάπτυξη, είναι ένα θέμα της προστασίας δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και να μπορέσουμε να έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία για να επιτύχουμε τους κλιματικούς στόχου που έχουμε θέσει στο Παρίσι. Αυτό είναι σε αδρές γραμμές ε, το μήνυμα που θα ήθελα να περάσουμε. Ξέρετε πώ λειτουργεί. Έχουμε έναν συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων στη συγκεκριμένη γνωμοδότηση αλλά ευχαρίστως ε, να ακούσω τις παρατηρήσεις σας για να βελτιώσω το κείμενο και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε κάτι το θετικό στο τέλος και πολύ σαφές να το υποβάλουμε στην Επιτροπή Μεταφορών για να τους πούμε ότι ναι μεν είναι δυναμικ... πολύ... μια πολύ δυναμική προσπάθεια στο πλαίσιο των ε, αγορών αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και όσον αφορά την περιβαλλοντική τύχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα έχω και συζητήσεις με τους κοιόδης εισηγητές για να έχουμε μια καλύτερη, μια καλύτερη έκθεση καλύτερη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο, να δώσω τώρα το λόγο στου σκιώδει εισηγητέ. Κύριο Δεμεσμάκερ, Προφανώ είστε ο πρώτο που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κανένα πρόβλημα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο γνωμοδότησής της. Πράγματι, έχουμε μεγάλες προσδοκίες σε σχέση με αυτά τα συνεργατικά FEE συστήματα μεταφορών. Είναι πολλά υποσχόμενα. Αυτά τα CITS, τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών, θα καταστήσουν τις μεταφορές μας πιο βιώσιμες, πιο αποτελεσματικές, πιο σίγουρες ε, λόγω της έρευνας και ανάπτυξης. Ο τομέας αυτός ε, προσελκύει πολλές επενδύσεις σε όλο τον κόσμο. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα σημαντικό μήνυμα για να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να πρωτοστατήσει. Στον τομέα αυτό η Φλάνδρα, που είναι και η περιφέρεια που εκπροσωπώ εγώ, ήδη συμμετέχει ενεργά σε αυτά τα ευφυή e e συστήματα μεταφορών, τα συνεργατικά, το Citrus, το, το European Citrus θα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα αυξήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα, θα μειώσει τις εκπομπές αερίων ε, και σε σχέση με την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων και θα βελτιωθεί και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Η συνάδελφος Σάλντε Μόζε μίλησε για το θέμα αυτό συζητούμε ε, και συνεργαζόμαστε με τις κάτω με τη Γαλλία, με το Ηνωμένο Βασίλειο για να υπάρξει ένα πιλωτικό πρόγραμμα που θα τονίσει ακριβώς τα στοιχεία αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα. Αυτό είναι το πρώτο και το πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρχει κάτι το ουδέτερο από τεχνολογικής απόψεως. Είμαστε υπέρ της τεχνολογικής ουδετερότητα. Όλα αυτά τα συστήματα μπορούν να συνεισφέρουν σε καλύτερη ποιότητα ε, του ατμοσφαιρικού αέρα, ε, βελτίωση της ενεργειακής μα αποδοτικότητας, αλλά πρέπει επίσης να σκεφτούμε και μακροπρόθεσμα, να σκεφτούμε τις δυνατότητες του συστήματος αυτού σε σχέση με τι δημόσιε μεταφορέ και με το συνδυασμό των ε, ιδιωτικών και των δημοσίων ε, ε, μέσων μεταφοράς. Πρέπει και τα ιδιωτικά οχήματα να μπορούν και εκείνα να συμμετέχουν σε αυτά τα συνεργατικά συστήματα μεταφορών. Το ζήτημα τώρα της ε, ευθύνης και των προ... της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ε, νομίζω ότι θα τα καλύψει η Επιτροπή Λίμπε, είναι και αυτά πολύ σημαντικά και σε σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα ήθελα πάντως να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και καλό σημείο αφετηρίας. Ένα μικρό πράγμα μόνο θα ήθελα να πω. Ε, πράγματι πρέπει να προσαρμοστεί το νομικό πλαίσιο, χρειάζεται ένα καλύτερο νομοθετικό πλαίσιο. Όμως υπάρχει ήδη μία οδηγία για τα ΕΦΗ e e αυτά συστήματα. Γι' αυτό πρέπει, πιστεύω, να την εκμεταλλευτούμε πλήρως. Και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Στρατηγική της αυτό προτείνει. Με αγωνία λοιπόν θα περιμένω τη συνεργασία με την εισηγήτρια ε, ώστε να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Κυρία Κονέτσνα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τη συναδελφό πολύ αξιόλογο το σχέδιο κειμένου. Περιέχει όλα όσα μας προβληματίζουν. Μπράβο που εμπλέκεται η Επιτροπή Περιβάλλοντος για τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και εμπλέκεται και στην προσπάθεια να μειωθούν οι βλαπτικές εκπομπές από τις μεταφορές και επίσης να προστατεύσουμε την υγεία μας από τις άλλες βλαπτικές ουσίες όπως το, το, τα, τα οξύδια του αζότου, τα άλλα σωματίδια, όλα αυτά θέλουμε να τα τυθασεύσουμε, να τα μειώσουμε στις πόλεις, ιδίω στις πόλεις. Και εκεί που πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο πώς θα μειωθούν όλα αυτά τα PM10, το PM5, όλα αυτά τα σωματίδια και μικροσωματίδια. způsobují a jsou karcinogenní a způsobují různé další zdravotní problémy. Takže já jsem moc ráda za to, jak je to... Όλα αυτά τα οποία μπαίνουν στον οργανισμό μας, όλα αυτά που είναι καρκινογόνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πρωτοπόρα σε αυτό το μέτωπο. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτά τα συστήματα μεταφορών. Αυτό το κάνουμε εμείς, θα το κάνει κάποιος άλλος αντί για μας. Ε, ε, Αυτό πρέπει να γίνει με αυτά τα ευφυή e συστήματα. Έχουμε περισσότερες δυνατότητες, να έχουμε περισσότερους πόρους σχετικά με αυτή την προσπάθεια και θα πρέπει να θεσπιστεί η κατάλληλη νομοθεσία. Οπότε θα πρέπει όλες αυτές οι ιδέες να είναι δυνατόν να υλοποιηθούν να μπορέσουμε να επικαιρώσουμε όλα τα εμπόδια που υπάρχουν στο κράτη-μέλη και αυτά τα συστήματα να δοκιμαστούν από κάθε κράτος. Πολλές φορές η νομοθεσία ε, είναι φραγμός στην ε, γρήγορη εφαρμογή ε, κάποιων ιδεών, κάποιων προτάσεων και πάμε σε τριετίες, πενταετίες καθυστέρησης. Και αυτό γιατί πολλά κρατημέλια δεν έχουν την νομοθεσία που προσφέρεται ούτως ώστε να προβούν σε αυτές τις καινοτόμες εφαρμογές. Εν κατακλείδη, έχω να σας πω ότι ναι, έχουμε τις κατάλληλες οδηγίες, όμως δεν γίνεται σωστή εφαρμογή τους. Άρα, να δώσουμε στα κρατημέλια τα κατάλληλα κίνητρα. Αλλιώς δεν ωφελούν τα νομοθετήματα. Θα πρέπει 25, 27, εν περιπτώσει, να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει, με, έρευνα, με, πρόσωπα, με, με εταιρείε. Αλλιώ θα μείνουν όλα αυτά νεκρογράμμα και θα είναι κρίμα. Že moc děkuji paní zpravodajce, για se συνεργασία spolupráci ε, e, σε σχέση με τις εξελίξεις και πάλι ευχαριστούμε την εισηγήτρια θα συνεργαστούμε μαζί της και ελπίζουμε ότι θα προσπάσουμε τελικά ένα σωστό, καλό, θετικό αποτέλεσμα Πρόεδρο ευχαριστούμε Επόμενος Κύριε Μιλέρα ευχαριστώ πολύ Εγώ δεν εκπροσωπώ το σκιώδη εισηγητή αλλά είναι τα προσωπικά μου σχόλια, προσωπικές μου παρατηρήσεις αυτές που θα σας αναφέρω σε ό,τι αφορά αυτή τη στρατηγική για τα ευφύ μεταφορικά συστήματα. Θεωρώ ότι είναι κάτι αναγκαίο και ιδίως ε, στην περίπτωση πόλεων που έχουμε κατάρρευση της κυκλοφορίας ε, με όλο και μεγαλύτερες ουρές ε, και μποτιλιαρίσματα που σίγουρα όλα αυτά επιβαρύνουν το περιβάλλον. Υπάρχουν δύο-τρία σημεία που θεωρώ ιδιαίτερο σημαντικά. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά ε, για την έκθεση αυτή πρωτοβουλία. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε ισχυρά επιχειρήματα. Έχει να κάνει σίγουρα το θέμα με την ε, πρότυπη των καταναλωτών και την προστασία των δεδομένων. Είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη αυτό. Και το άλλο σημαντικό για μένα είναι ο ρόλος ε, των πόλεων, των δήμων και κοινοτήτων, ιδίως ό,τι αφορά τις συγκοινωνίες. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε τον, το σχεδιασμό των ε, συνεργατικών αυτών ε, μεταφορών και το τρίτο που θέλω να αναφέρω είναι το δυναμικό, οι δυνατότητες ε, που προσφέρουν αυτές οι συνδυασμένες μεταφορές για μεγαλύτερη αποδοχή από πλευράς καταναλωτών. Τα ηλεκτρικά οχήματα ε, θα έχουμε γι' αυτά σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες ε, και ακόμη και για τους σταθμούς ε, φόρτισης. Ε, όλα αυτά θα βοηθήσουν τη μεγαλύτερη αποδοχή, επαναλαμβάνω, εκ μέρους των καταναλωτών. Θα καταθέσω και σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τώρα εκ μέρου τη Κομισιόν, ο κ. Βάντεν Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που μας καλέσατε και μας δώσατε την ευκαιρία να σχολιάσουμε τα της στρατηγικής αυτής. Ευχαριστούμε που μας στηρίζετε γιατί το πώ θα αυτά τα συστήματα, πώ θα εφαρμοστούν, έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα όσον αφορά τι οδικέ μεταφορέ. Αυτά τα δύο είναι ελληνέντετα, γιατί όταν έχουν περφορτωμένο οδικό δίκτυο, ένα μικρό περιστατικό φέρνει χάο και βλάπτει και το περιβάλλον. Ε, Επομένω, και εμεί ακράδαντα πιστεύουμε ότι τα σχετικά συστήματα βοηθούν και για την ροή τη ε, κυκλοφορία, αλλά και ακριβώς όπως είπατε, έτσι έρχεται να συνδυαστεί η μεταφορά ε, η οδική με άλλους τρόπους ε, μεταφοράς. Και το ισχύει για χώρους Ε, επίσης σας τονίζω πως τονίζουμε ότι ήδη υπάρχει υποστήριξη για αυτή την ιδέα πριν από δύο εβδομάδες. Στο Ταλίν γιορτάσαμε Ε, την διεύρυνση ε, αυτού του συνόλου κρατών που ασχολούνται με αυτό το μέτωπο των 16 εκατομμυρίων με τις τρίτες χώρες και είπαμε ότι αυτό πρόκειται να ε, ωφελήσει όλου του είδους τα οχήματα, όλου, πολλούς κλάδους, όλους τους χρήστες τέλο πάντων του, του οδικού δικτύου. Και αυτό έχει σχέση και με την επίδειξη του στόχου του 2029, οπότε έχουμε δεσμευτεί και οι αρχές, αλλά και ε, ο επαγγελματικό κλάδος ότι είναι πλεονέκτημα αυτό το οποίο έχει η Ευρώπη με το να είναι πρωτοπόρα σε αυτό το μέτωπο. Κυρία Σαλντεμόσε, θέλετε να δευτερολογήσετε στα δανέζικα. Ναι, ναι. Σύντομα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους Πλησέτε τη βοήθειά του για αυτό το σχέδιο κειμένο. Νομίζω ότι σύντομα είπανε πάρα πολύ εύστοχα πράγματα, βελτιώνουν το κείμενο και είναι υπόμονο περιμένω συνεχιστή συνεργασία μας. Πρόεδρος. 1η Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία στις 11 η ώρα για τις τροπολογίες. Ψηφίζουμε 24 Ιανουαρίου στην ΕΝΒΗ και στην ΤΡΑΝΣ τον Φεβρουάριο. Και τώρα προχωρούμε 106 όσον αφορά το φωσφορούχα στο κρέας. Κύριε Σολτεμός και κύριο Στάση έχουν αναλάβει αυτό το κείμενο. Κύριε Σολτεμός πρώτη θα μας τα πει. Σας ευχαριστώ. Άλλο θέμα τώρα, Πρόεδρε. Τελείω διαφορετικό. Πρώτη τη σχετική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τροποποιεί τον ε, κανονισμό 1063 του 2008 και αφορά την χρήση διαφόρων φωσφορικών ουσιών όσον αφορά το κατεψυγμένο κρέας ε, που χρησιμοποιείται, αξιοποιείται τέλο πάντων κάθετα όπως ο γύρος Φερρυπίν, το σαβαρμά κλπ. Έχουμε αυτά τα φωσφορούχα τα οποία κατά κάποιο τρόπο είναι φυσικέ ουσίες. Ουδές κίνδυνο για το πεπτικό. Øh, er er Οπότε έχουμε από την άλλη μεριά όμω πρόβλημα από τα τεχνητά, τεχνητές ουσίε ουσίες που υπάρχουν. Οπότε ε, υπάρχουν τέτοια πρόσθετα στα είδη διατροφής. Οπότε εδώ έχουμε μια σειρά επιφυλάξεων ανησυχιών από πλευρά της επιστημονικής κοινότητας. Και λέμε ότι η χρήση αυτών των επικίνδυνων ουσιών μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο για τις καρδιογγειακές παθήσεις. Στην ΕΦΣΑ αυτό αποτελεί υπόθεση προτεραιότητος. Και η ΕΦΣΑ τώρα αξιολογεί το τι συμβαίνει ακριβώς με αυτές τις επικίνδυνες φωσφορούχες ουσίες. Τέλος του 18 θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η εξέλιξη. Επομένως, τα φωσφορούχα τα φυσικά εγκλίνουν κανένα κίνδυνο, ενώ αντιθέτως αυτό ισχύει για τα, για τα τέλος πάντων. Οπότε είπαμε προσοχή ε, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε πλην, πριν η ΕΦΣΑ ε, παραδώσει την αξιολόγησή της ε, τα τέλη του επομένου έτους. Βεβαίως και είναι σοβαρό πρόβλημα οι καρδιαγγικές παθήσεις στην Ευρώπη. Οπότε να μην τα κάνουμε τα πράγματα ακόμα χειρότερα με αυτές τις τεχνητές φωσφορικές ουσίες όσον αφορά αυτά που τρώμε. Ε, βέβαια, ε, φυσικά και δεν τρώει κάθε μέρα κανείς ε, αυτού του είδους της λιχουδιές, αλλά όμως είναι σημαντική η κατανάλωση, οπότε αυτό είναι μια μεταβλητή που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και δεν είναι θέμα μόνο καρδιακές παθήσεις, υπάρχει και ζήτημα νεφρολογικό. Ε, επομένως όλα αυτά πρέπει να προσέξουμε σε σχέση με τα κρέατα. Θέλουν και άλλοι συνάδελφοι να προσθέσουν τα επιχειρηματά τους. Πάντως, επί τη βάση όλων σας ανέπτυξα, θα πρέπει να μην προχωρήσουμε στην τροποποίηση του κανονισμού. Να περιμένουμε την έκθεση της ΕΦΣΑ και να δούμε αν πραγματικά ενεδρεύουν εδώ κίνδυνοι. Πάντως εμείς βάσιμα ανησυχούμε όσον αφορά τα μη φυσικά φωσφορούχα. Άρα προτείνουμε όχι στην πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θεωρούμε ότι τα φωσφορούχα αυτά πρέπει να μπουν στο δεύτερο και τρίτο παράρτημα με τις σχετικές ουσίες. Άρα θα πρέπει εδώ να ισχύσει η αρχή της ε, επιφύλαξης γιατί υπάρχουν ενδεχόμενα συνέπειες της χρήσης αυτών των ουσιών επί της υγείας μας. Άρα, αναμονή μέχρι να γνωμοδοτήσει η ΕΦΣΑ. Διότι η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η υγεία του κόσμου. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την ε, ένσταση. Φαντάζομαι την έχουμε πρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις ενστάσεις μας, αλλά ο στόχος μας είναι το συμφέρον των Ευρωπαίων και ο συνάδελφος Μπανιστάς από τους Πρασίνους πρόκειται επίσης να παρουσιάσει διάφορα επιχείρηματα και έτσι θα δικαιολογήσει και εκείνος αυτή την πρόταση ε, ένστασης. Δεν πιστεύω ότι η Κομισιόν ε, θα ενοχληθεί αν προβάλλουμε αντίρρηση. Τέλος πάντων, και εμείς καταναλωτές είμαστε όλοι προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την υγεία ε, ευεξία των καταναλωτών. Ο συνάδελφος Μπάρτ Πέρτ Στάς. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Σάλντε Μόζε. Και όπως είπε και η ίδια μόλις πριν, μιλάμε εδώ για τα φωσφορικά τα οποία προστίθενται στα ε, κρέατα ε, που καταναλώνουμε με τη μορφή γύρου σε κάθε σούγκλες. Ε. Έχουμε λοιπόν τους ε, τις ουσίες τα D3 πολυφωσφορικά άλλα, τα ε338, 452. Υπάρχει το άρθρο 6 του κανονισμού 1333-2008 και πρέπει να γίνονται σεβαστά συγκεκριμένα κριτήρια για, για τα πρόσθετα τροφίμων. Δεν πρέπει να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών, για τη υγεία δεν πρέπει να υπάρχει ένα, μια άλλη τεχνολογική δυνατότητα και βέβαια δεν θα πρέπει να παραπλανάται ο καταναλωτής. Στο ψήφισμα το οποίο έχουμε και το οποίο θα τεθεί αύριο σε ψηφοφορία, εμείς έχουμε προβάλει μια σειρά από επιχειρήματα και λέμε ότι αυτά τα κριτήρια δεν γίνονται σεβαστά. Είπε και η κυρία Σάλντε Μόζε ότι πράγματι Υπάρχουν αμφιβολίες και από επιστημονικής ε, πλευράς, δεν συμφωνούν μεταξύ τους οι επιστήμονες, δεν ξέρω κατά πόσο είναι επιβλαβή αυτά τα λατά ή όχι για την ε, ανθρώπινη. Για άλλε ε, μελέτες δείχνουν ότι για το καρδιακιακό σύστημα δεν είναι καλά αυτά τα φωσφορικά λατά και η ΕΦΣΑ τα λέει κάπως συγκεχημένα στη μελέτη. Γι' αυτό καλό είναι να υπάρξει δεύτερη μελέτη, την οποία θα την έχουμε μέχρι τέλος του 2018. Μέχρι να έχουμε αυτή τη μελέτη, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε την Κομισιόν και να δεχθούμε την πρότασή της για αυτά τα τεχνικά, τεχνητά φωσφορικά Η προσθήκη δε τέτοιων ουσιών μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή. Αν προσθέσουμε φωσφορικά άλατα, αυτό μπορεί να το κάνει κάποιος απατεώνας. Και προσθέτει ίσως και περισσότερο νερό στο κρέας που πουλιέται ε, με στην τιμή του κρέατος τελικά το νερό για τον καταναλωτή. Μπορεί αυτό να μην βλάπτει την υγεία του καταναλωτή, πάντως θεωρώ ότι αυτό είναι απάτη και παραπλάνηση του καταναλωτή. Επίσης, από όλες ε, τις επιστημονικές μελέτες ε, αποδεικνύεται ότι δεν είναι αυτή η πρακτική απαραίτητη, γι' υπάρχουν και άλλες εναλλακτικέ. άρα ούτε αυτό το κριτήριο γίνεται σεβαστό, το κριτήριο του άρθρου 6, δηλαδή του κανονισμού 1333 του 2008 και τέλος αυτό το είδος του κρέατος, οι γύροι αυτή, χρησιμοποιούνται ε, σε μικρά, μάλλον πολλούνται σε μικρά καταστήματα, κεμπάμπ, fast food ουσιαστικά και δεν υπάρχει και επισήμανση του προϊόντος. Δεν ενημερώνει το καταναλωτής, δεν ξέρει τι καταναλώνει, τι υπάρχει μέσα στην πίτα που τρώει, μέσα στο πιάτο που έχει παραγγείλει να φάει. Είναι πολύ δύσκολο με τα σκευάσματα αυτά κρέαντος Πολλές συζητήσεις ε, έχουν ξεκινήσει και ομοφωνία μεταξύ των υπηρεσιών επιθεώρησης δεν υπάρχει. Δύσκολο λοιπόν και περίεργο είναι πράγματα που ήδη τώρα δυσκολευόμαστε να ελέγξουμε, να είμαστε έτοιμοι να τα δεχθούμε. Αντί λοιπόν να νομιμοποιήσουμε τις πρακτικές αυτές, νομίζω ότι πρέπει να εντείνουμε τους ελέγχους στα κράτη-μέλη και έχουμε την νομοθεσία που ήδη υφίσταται και αυτή πρέπει να ε, εφαρμοστεί και να ενισχυθούν οι έλεγχοι ώστε οι καταναλωτές να μην εξαπατώνται. Αυτά. Πιστεύω ότι η κυρία Σαλτεμόζε σας παρουσίασε όπως και εγώ αρκετά επιχειρήματα που βασίζονται στο άρθρο 6, όπως είπα, του κανονισμού του σχετικού, ώστε να πιστείτε κι εσείς ότι η Κομισιόν δεν ε, θα πρέπει να ε, επιτρέψει την ε, χρήση αυτών των φωσφορικών αλάτων. Ο Ιβο Μπέλετ. Εντάξει, την ίδια πολιτική οικογένεια με τη συνάδελφο. Θα είμαι σύντομος. Να πω και εγώ δύο λόγια εκ μέρους της Ρενάτε Ζόμερ που ακόμη είναι στο δρόμο, γιατί έρχεται Βρυξέλλες, δεν έχει φτάσει ακόμη. Να προσθέσουμε λοιπόν ε, κάποια άλλα επιχειρήματα σχέση με αυτά που έχουν ακουστεί ήδη. κατάρχα αρνητικέ ε, δυνητικά ε, επιπτώσει στην υγεία, τα φωσφορικά αυτά άλατα. Υπάρχει μία αναφορά από την ΕΦΣΑ από το 2013 που λέει ότι δεν έχουν εντελώς πιστικές ε, αποδείξεις ε, οι σχετικές μελέτες για το κατά πόσο είναι επιβλαβή αυτά τα, ε, αυτές οι ουσίες. Το δεύτερο επιχείρημα ότι δεν υπάρχει τεχνολογική ανάγκη για τη χρήση αυτών των φυσορικών αλάτων. Είναι σαφές με βάση εμπειρογνώμονες ότι έχουν σταθεροποιητικό, συγκολητικό αποτέλεσμα ή συνδετικό αυτά τα φωσφορικά άλατα γιατί αλλιώς ε, δεν συγκρατούν, δεν συγκρατείται το κρέας ε, στους, στις σούβλες αυτές. Ε, αυτό λένε οι εμπειρογνώμονες, άρα υπάρχουν και τεχνολογικά επιχειρήματα για τη χρήση των φωσφορικών αυτών Αλλά Ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι η χρήση των φωσφορικών αυτών είναι, λέγεται, παραπλανητική, λόγω των ιδιωτήτων τους που διατηρούν ε, το, το νερό. Φυσικά δεν θέλουμε να υπάρχει τέτοιου είδους εξαπάτηση. Αυτές οι σούβλες, αυτοί οι γύροι, ε, ποτέ πρέπει να καταναλώνονται εκτός σπιτιού. Ε, ακόμη και στα fast food που αγοράζονται κατεψυγμένα ε, μπιφτέκια, βλέπουν το περιεχόμενο του νερού, την περιεκτικότητα του κρέατος σε νερό. Αυτό το ε, επιβάλλει ο κανονισμός το 2011. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα με την περιεκτικότητα σε νερό. Και ένα τελευταίο επιχείρημα ότι δεν υπάρχει ενημέρωση των καταναλωτών για την ε, περιεκτικότητα των σκευασμάτων αυτών σε φωσφορικά άλετα. Στο άρθρο 44 τα κράτη-μέλη έχουν την ευχαίρεια να ε, υιοθετήσουν εθνικές διατάξεις για τα προσκευασμένα αυτά προϊόντα. Άρα, κατ' εμάς, ε, η πρόταση της Κομισιόν Απλά διευκρινίζει κάποια πράγματα για αυτά τα κατεψυγμένα, στους κατεψυγμένους γύρους, ε, ότι μπορούν να περιέχουν τους ίδιου, τα ίδια, την ίδια ποσότητα ε, φωσφορικών αλάτων που έχει εγκριθεί για άλλα προϊόντα ε, εδώ και καιρό. που χρησιμοποιούνται σε ψητοπολία. Ευχαριστώ. Thank you very much. Is there any, uh, other... Ευχαριστώ. Υπάρχει κανένας άλλος συνάδελφος που θα θέλει να πάρει το λόγο. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια ερώτηση. Αυτό βασίζεται στο ε, κέντρο τεχνολογικών ερευνών που όντως δημοσίευσε αυτές τις ανησυχίες, από πού προκύπτουν αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει τέτοια συζήτηση αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, τελικά τι θα γίνει στις Ηνωμένε Πολιτείε τα φωσφορικά άλατα σε τέτοιου είδους κρέας θα ε, απαγορευτεί. Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Κυρία Κονέτσινα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω ορισμένα πράγματα εκ μέρους της ομάδας μου που υποστηρίζει την αντίρρηση αυτή. Το θέμα δεν είναι κατά πόσο τα κεμπαμπτζίδικα θα έχουν ε, τεράστιες ποσότητες ε, κρέατος ε, γύρω από μία σούβλα που γυρίζει γύρω-γύρω κάθετα. Ε, το θέμα είναι η προστασία των καταναλωτών. Αυτό μας ενδιαφέρει. Όχι να κοιτάμε τα κεμπαμπτζίδικα, να κοιτάμε τους ε, καταναλωτές και την υγεία τους. Η ΕΦΣΑ αυτή τη στιγμή εξετάζει εκ νέου την ασφάλεια των φωσφορικών αλάτων ε, ως ε, πρόσθετων τροφίμων. Κάποια στιγμή, κατά τη τέρια του 2018, θα έχουμε τα αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε αρκετό, αρκετά μεγάλο κίνητρο όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μην λάβουμε ε, βήματα τα οποία δεν θα λαμβάνουν αυτό υπόψη. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τη χρήση των ε, αλάτων αυτών ε, στα, στο κρέας εφόσον υπάρχει μια μελέτη στο πλαίσιο της ΕΦΣΑ, γιατί να μην περιμένουμε. Γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε υπευθύνω να δηλώσουμε ότι η πρόληψη είναι η προστιθέμενη αξία των, της ευρωπαϊκής πολιτικής, ώστε οι ευρωπαϊκοί οι ευρωπαίοι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς. Του είπε κάποιος συνάδελφος στην Τσεχία υπάρχει πάρα πολύ απάτη την οποία προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε. Ε, χρησιμοποιούνται κάποιες απατηλές πρακτικές με τη χρήση ουσιών ε, και επιπλέον ε, ύδατος στο κρέας για να αυξηθεί το βάρος του κρέατος αντί να ε, βοηθούμε τα κράτη-μέλη στην καταπολέμηση αυτών των πρακτικών εξακολουθούμε να ανοίγουμε πόρτες στη χρήση των πρακτικών αυτών και αυτό δεν θα πρέπει καθόλου να το κάνουμε κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω την υποστήριξή σας στην αντίρρηση αυτή εκ μέρους της ομάδας μου Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για την υποστήριξη αυτή και αν δεν ασχολούμαστε τόσο με τη λειτουργία των ε, ε, κεπαπτζίδικων αλλά με τη δημόσια υγεία, νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλη, όλη την αντίρρηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μιλάμε τώρα για τα φωσφορικά άλατα στις, ε, στο, στο, στο κατεψυγμένο κρέας που τοποθετείται σε σούβλα. Ε, πρόκειται λοιπόν για μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση. Ε, η αίτηση εξέτασης της, του κρέατος αυτού ελήφθη το 2016 και συζητήθηκε πάρα πολύ εντατικά με την ομάδα εργασίας κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων για τα πρόσθετα τροφίμων συγκεκριμένα σε σχέση με το κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμπερίληψη και τη χρήση ε, των ε, προσθέτων τροφίμων ε, στο πλαίσιο της υφισταμένης νομοθεσίας. Τα κράτη-μέλη λοιπόν συμμετείχαν βεβαίως στην διαδικασία αυτή. Βάσει του άρθρου 6.333 του 2008 μπορεί ένα πρόσθετο να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των, της Ένωσης μόνο αν πληρούνται κάποιες Πρώτον, βάσει επιστημονικών ε, αποδεικτικών στοιχείων ε, και αν δεν δημιουργεί, δεν αποτελεί απειλή στο επίπεδο και τη συγκέντρωση χρήσης ε, στους πολίτες. Επίσης, αν υπάρχει μια τεχνολογική ανάγκη η οποία δεν μπορεί με άλλον οικονομικό ή ε, τεχνολογικός πρακτικό τρόπο να ε, επιτευχθεί, αν δεν παραπλανεί ε, τους πολίτες και επίσης πρέπει τα πρόσθετα τροφίμων να έχει κάποιο όφελος και για τους πολίτες και για να μπορεί επίσης να βοηθήσει ...στην επίτευξη των στόχων που ανέφερα παραπάνω. Για να μπω τώρα λίγο σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες όλων αυτών των προϋποθέσεων, καταρχάς το θέμα της ασφάλειας των φωσφορικών αλάτων αξιολογήθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή για τα Τρόφιμα το 1991 και μία, ετήσια προς, μία ημερήσια πρό, πρόσληψη 17 ε, μιλιγκράμμ ε, ορίστηκε Επίσης ε, αδειοδοτήθηκε σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως προϊόντα κρέατος και κάποια παρασκευάσματα κρέατος ε, και φυσικά και στις ε, κάθετες σούβλες όπου υπάρχει κατεψυγμένο κρέας και είχαμε, είχε αποφασιστεί τότε ότι δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ως προς τη συνολική έκθεση στα φωσφορικά άλατα. Κατόπιν αιτήματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι το οποίο αναφέρθηκε στη συζήτηση, η ΕΦΣΑ το 2013 αξιολόγησε ε, την αναθεώρηση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με τα φωσφορικά αλάτα και τη χρήση τους. Η ΕΦΣΑ όμως δεν ε, ε, αμφισβήτησε την προηγούμενη γνωμοδότηση και τα συμπεράσματα της Επιστημονικής Επιτροπής για τα πρόσθετα τροφίμων που είχε ορίσει αυτήν την ημερήσια πρόσληψη ε, και τα επίπεδα αυτής και που τότε θεωρήθηκαν ασφαλή. Κάτι ακόμη να σας πω, εν είδη πληροφορίας, γίνεται ένα πρόγραμμα εκ νέου αξιολόγησης για τα πρόσθετα τροφίμων, όχι μόνο για τα φωσφορικά άλατα. Αλλά για το επίπεδο της χρήσης των προσθέτων τροφίμων, μέχρι το τέλος του 2018 πρέπει να έχει γίνει ε, αυτή η εκ νέου αξιολόγηση των φωσφορικών αλάτων. Στο πλαίσιο αυτό, τα πιο σημαντικά και ενημερωμένα επιστημονικά δεδομένα θα αξιολογηθούν από την ΕΦΣΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως παρακολουθεί την κατάσταση εκ του και αν υπάρξει ε, λόγος θα εξετάσει το ενδεχόμενο ύπαρξης ε, μέτρων ε, ε, κατόπιν δημοσίευση των πορισμάτων της μελέτης αυτής. Ε, αυτή τη στιγμή ε, δημοσιευθεί η μελέτη της ΕΕΠΣΑ, ε, θα το κάνουμε αυτό. Μέχρι τότε εξακολουθούν να ισχύουν τα επίπεδα που, είχαν οριστεί, που είχαν οριστεί στο παρελθόν και που ισχύουν και τώρα. Όσον αφορά τώρα την τεχνολογική ανάγκη. Η τεχνολογική ανάγκη αναγνωρίστηκε για κάποιες σούβλες κρεάτων, όπως αναφέρεται στο σχέδιο κανονισμού, τα φωσφορικά άλατα είναι απαραίτητα για τη σταθεροποίηση των κρεάτων και ε, προκειμένου να παραμείνουν να παραμείνει το κρέας ε, ενωμένο, για να υπάρχει ομοιογενής ψήξη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος ε, ε, διαφορετικής μεταχείρισης του κρέατος που ήδη αποτελεί ένα κίνδυνο για την υγεία. Δεν υπήρξαν άλλες εναλλακτικές πρακτικές που να εντοπίστηκαν τότε. Επίσης υπήρχε η απέτηση της μη παραπλάνησης του ε, πολίτη. Όταν μιλάμε για τον τομέα επιχείρηση προς επιχείρηση, το επιπλέον νερό πρέπει να προστίθεται ε, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Όσον αφορά τώρα ε, το, κρέα, το, το νερό στον οπό κρέας, τότε είχαμε αποφασίσει ότι πρέπει όταν υπάρχει φωσφορικό άλας να μην υπάρχει επιπλέον νερό, δεν χρειάζεται να υπάρχει επιπλέον ε, ε, νερό, οπότε ως επιπλέον ε, ε, πληροφορία, τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα υπό την τρέχουσα νομοθεσία να, υπάρξουν, ε, να ορίσουν επιπλέον εθνικά μέτρα ε, για ενημέρωση των πολιτών και για, το προσυσκευασμένο, και για τα προσυσκευασμένα γεύματα. Όσον αφορά τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές, τα φωσφορικά άλατα βοηθούν την κατασκευή και την επεξεργασία κάποιων κρεάτων σε κάθετες σούβλες, ε, ε, επομένως ε, πληρούν πλήρως τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν είναι της απόψεως ότι το σχέδιο κανονισμού πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του σχετικού κανονισμού 1333 του 2008. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ βεβαίως και εγώ. Η κυρία Σάλντε για να συνοψίσει. Και μετά ο κύριος Στάσης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να επαναλάβω ότι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε αυτή την πρόταση για μια αντίρρηση, για την υποβολή αντίρρησης, είναι γιατί δεν θεωρούμε να περιμένουμε άλλο. Η ΕΦΣΑ θεωρεί ότι είναι υψηλή προτεραιότητα σε αυτό το θέμα και μα υποσχέθηκε ότι θα έχει τελειώσει την αναθεώρησή τη εντό ενό έτου. Και θεωρούμε ότι εφόσον υπάρχουν ήδη κάποιε συζητήσει ε, ε, στον επιστημονικό χώρο σε σχέση με τον κίνδυνο αυτών των προσθέτων τροφίμων, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να περιμένουμε και να δούμε τι θα μας πει η ΕΦΣΑ. Καλό είναι να περιμένουμε. Ε, το έχουν ε, ε, πλέον στο πρόγραμμα εδώ και ένα χρόνο, μάλλον μπορούμε να περιμένουμε ένα χρόνο ακόμη πριν πάρουμε μια απόφαση. Νομίζω ότι είναι ένα βασικό επιχείρημα αυτό. Να περιμένουμε, αυτή τη στιγμή η ΕΦΣΑ θα ε, τελειώσει την έρευνά τη, την αναθεώρησή τη. Είναι κρίμα να λέμε, είναι, είναι μάλλον ανόητο να πούμε ναι στην αλλαγή αυτή του κανονισμού αντί να περιμένουμε αυτόν τον επιπλέον χρόνο. Ε, και έτσι θα μπορέσουμε άλλωστε να προστατεύσουμε και καλύτερα του καταναλωτέ. Αυτό είναι το κύριο μα επιχείρημα. Δεν ξέρω τι κάνω στι ΗΠΑ, κυρία Πρόεδρε. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες επιστημονικές ανησυχίες, ε, αλλά δεν ξέρω από νομοθετική απόψεω τι έχουν σκοπό να κάνουν. Πάντω, επειδή εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το ύψιστο επίπεδο ασφάλεια τροφίμων, ε, α μην ασχολούμαστε με τι ΗΠΑ, ασχολούμαστε περισσότερο με το τι γίνεται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κύριο Στά, συμφωνώ 100% με την συνάδελφο. Και να σα πω, κύριε Σούμερ Βάρκε, κύριε Μπέλετ, τα εξή ότι όσον αφορά την μελέτη της ΕΦΣΑ δεν έχουν υπάρξει προς το παρόν κάποια συμπεράσματα ασφαλή όσον αφορά τη υγεία Αλλά η ΕΦΣΑ θέλει να κάνει μια αξιολόγηση εκ νέου μέχρι το τέλος του επόμενου έτους τόσο τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα. Ακριβώς όπως τα είπε η κυρία Σόλτεμόζε. Αυτά και από πλευράς ε, τεχνικής τεχνολογίας, η ίδια η ΕΦΣΑ πάντως, αυτό το οποίο διακηρύσει ε, είναι ως επιχείρημα ότι το κεμπάπ το οποίο πωλείται δεν περιέχει τεχνητά φωσφορούχα. Επομένως, από πλευράς τεχνικής, τεχνολογικής, ε, είναι δυνατόν να προωθηθεί, να υπάρξει, να παραχθεί το προϊόν χωρίς αυτές τις ουσίες. Η Επιτροπή πιστεύει ακράδαντα ότι δεν πρόκειται για ουσίες που παχαίνουν. Ούτε πολλά κανείς φύγει για μεταξύ κορδέλες. Ε, τελικά εμείς λάβαμε υπόψη τα στοιχεία που έχουμε εκεί, από ό,τι φαίνεται ότι θα πρέπει να το ψάξουμε περισσότερο. Δεν υπάρχουν μέχρι τώρα οριστικά συμπεράσματα. Γι' αυτό σας λέω. Να απορρίψουμε την πρόταση της Επιτροπής. Να περιμένουμε την ΕΦΣΑ να ολοκληρώσει την αξιολόγηση και μετά να αποφασίσουμε. επιφέρουν αυτό που είπε η Το 2013-2014 είχαμε κάποιες μελέτες, είχαν δημοσιευθεί αφού η ΕΦΣΑ έκανε την πρώτη αξιολόγηση, οπότε και η επιρροή στην Αμερικανική νομοθεσία βέβαια δεν είναι γνωστή. Εμείς πάντως αρχίσουμε αυτή την ώρα και φυσικά και πρόκειται να επικοινωνήσουμε σχετικώ μαζί σας. Να δούμε τι θα κάνουν οι Αμερικανοί. Ελπίζουμε να λάβουν υπόψη και αυτή την αξιολόγηση της ε, ΕΦΣΑ. Αύριο θα ψηφίσει η Επιτροπή μας επ' αυτού στη Διαλόμελια. Εάν εγκριθεί εδώ το κείμενο θα πάει τον Δεκέμβριο. Και τώρα προχωρούμε. Έχουμε την ε, συμφωνία, τη συνθήκη τέλο πάντων με την Ελβετία. σύνδεση του αίτιας των Ελβετών με το δικό μας αίτιας. Πολύ συμπαθητική αυτή η εξέλιξη. Ο κύριος Μπέλετ θα λάβει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε και πάλι. Ναι, ναι, ο κύριος Φιέλνερ που το έχει αναλάβει μου ζήτησε εκ μέρους του να πω δύο λόγια. Γιατί είμαι εξοικειωμένος με το θέμα Οπότε με τα χαράς να το αντικαταστήσουμε μια που πρόκειται για ένα ζήτημα ε, για το οποίο έχουμε ε, καταβάλει μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Ελβετία που άρχισαν πριν από έξι χρόνια. Οπότε τώρα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της υπόθεσης αυτής της διαδρομής, αυτών των διαπραγματεύσεων και βέβαια είμαστε υπέρ του να ολοκληρωθούν το Συμβούλιο ήδη απεφάσισε και έδωσε το πράσινο φω για αυτέ τι διαπραγματεύσει μεταξύ ΕΕ και Ελβετία, να συνδεθούν αυτά τα δύο συστήματα εκπομπών, τα δύο ETS. Ε, φυσικά και το ελβετικό σύστημα είναι πιο μικρό από το δικό μας και βέβαια εμεί ως ευρωβουλευτέ θα πρέπει και εμεί με τη σειρά να δώσουμε το πράσινο φω. Ε, δηλαδή αναμένεται από εμά να πούμε ένα ναι ή ένα όχι. Δεν είναι θέμα ψηφισμάτων και άλλων κειμένων. Το ETS ήδη έχει περάσει από τροποποιήσεις τελευταία, χρόνια, τελευταίους μήνες και κυρία Πρόεδρε, υπό τη δική σας Προεδρία έχουμε συζητήσει συμφωνώντας ότι η πολιτική ακρογωνία λίθο της πολιτικής της Ένωσης βασικό εργαλείο για να μειώσουμε τις εκπομπές αυτές που έχουν σχέση με το φαινόμενο θερμοκηπίου. Οπότε η σύνδεση του συστήματός μας με άλλα συστήματα μέσα στον κόσμο. Α, το τώρα που ξεκινάμε με την ε, Ελβετία. Τα είπαμε και πριν από δύο εβδομάδες στην συνάντηση της Βόνης για την αλλαγή του κλίματος. Είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το βήμα όσον αφορά να έχουμε ένα πραγματικά παγκόσμιο σύστημα ETS. Ε να μην μείνει αυτό ένα όνειρο, να γίνει πραγματικότητα. Να γίνει πραγματικότητα τα μέσα ομενά χρόνια. Όχι δεκαετίες, τέλος πάντων η σύνδεση των δύο ETS ε του μεγάλου του δικού μας και του μικρότερου ελβετικού δημιουργεί μεγαλύτερη αγορά και δίνει περισσότερες δυνατότητες για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών. αυτό φυσικά έχει σχέση με την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Να δούμε τι θα γίνει και με άλλους στην παγκοσμία σκηνή να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας. Ε, να, τους δίνετε τώρα ευκαιρία να δουν το πώς τα συνδυασμένα συστήματα μπορούν να αποδώσουν. Α, αυτά προτείνει και ο εισηγητής. Αύριο να επιψηφίσετε το κείμενό του. A large majority of support in, in, this, uh, in this chamber. Thanks. Thank you very much. Ευχαριστούμε. Ναι, πράγματι. είναι πολύ σημαντικό για τη στρατηγική αποστολή τη Ευρωπαϊκή. Ένωση. να πείσουμε να ακολουθήσουν και άλλοι την άποψη που έχουμε σε σχέση με την εφαρμογή του συστήματο ETS και το όραμά μα. Είναι πολύ ευτυχέ το γεγονό ότι η Ελβετία συμμερίζεται το δικό μας όραμα, από ό,τι φαίνεται. Πρέ... Στρέφουμε στους σκιώδες συζητητές. Ποιος παγνιό είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως πολύ σωστά μας πενθύμισε ο κύριος Μπέλετ, εξόμως του εισηγητή, επειδή έχουμε το κατεπήγον κλιματικής ε, αλλαγής, ε, θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις συμμαχίες μας ε, σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο και να έχουμε συνδυασμένα συστήματα ανταλλαγής δικαιωμάτων εκπομπών. Το 2019 θα προσθεθεί η Ελβετία. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ένα τέλειο παράδειγμα αυτής της νέας συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνδέσει την αγορά της, τη μεγαλύτερη, σε μία τρίτη χώρα. Και το 2019 συμμετέχονται στην αγορά ETS Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν επομένως να χρησιμοποιούν δικαιώματα από το ελβετικό σύστημα και αντιστρόφως. Αυτή η διασύνδεση λοιπόν θα ενισχύσει την ε, ε, χρησιμοποίηση των ε, δύο συστημάτων και ελπίζω να δημιουργηθεί μια στέρεη αγορά Εμπόρια δικαιωμάτων άνθρακα. Εκ μέρους ομάδος μου είμαι υπέρ της σύναψης της συμφωνίας. Σε ό,τι αφορά όμως τον τύπο, θα θέλαμε να είχαμε περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της συμφωνίας. Στο μέλλον λοιπόν θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο διαφανής όταν εκπονεί και συνάπτει ανάλογες συμφωνίες. Αυτά είχα να πω αγαπητοί πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι εκ μέρους της ομάδας μα Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Ε, κυρία να έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, και εμείς καλωσορίζουμε τη σύναψη της συμφωνίας αυτής, αν και βλέπουμε λίγο διαφορετικά το ETS σε σχέση με τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου. Πάντως, είναι καλό να υπάρχει ένα παγκόσμιο σύστημα, να προσπαθούμε να ε, εφαρμόσουμε ε, ένα παγκόσμιο σύστημα, γιατί μόνο εντός Ένωση ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να φέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε ένα μεγάλο άλμα πριν από μερικές εβδομάδες από κοινού με το Συμβούλιο και τώρα έχουμε κάτι να προσφέρουμε στους εταίρους μας. Έχουμε μια λύση να τους προσφέρουμε. Και πρέπει να υποστηρίξουμε οποιονδήποτε θέλει να έρθει στη δική μας, ε, στο δικό μας στρατόπεδο των εισαγωγικών. Ελπίζω σε κάποια χρόνια και όχι σε κάποιες δεκαετίες να μπορέσουμε να έχουμε ένα σύστημα πραγματικά παγκόσμιο. Τώρα, αν έχουμε ένα καλό σύστημα εδώ, σε αυτή την ε, περιοχή του κόσμου. Δεν θέλουμε να υπάρχει διαρροή άνθρακα σε άλλα μέρη του κόσμου. Εξού και πρέπει να συνάψουμε συμφωνίες με τρίτες χώρες, όπως η Κίνα για παράδειγμα, ή άλλους μεγάλους πρωταγωνιστές. Αν θέλουμε να είναι λειτουργικό μάλλον αυτό το σύστημα και αν θέλουμε να αποκομίσουμε τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη από αυτό το σύστημα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μείωση των εκπομπών δεξιδίου του άνθρακα, και αν θέλουμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας ε, μετά την διάσκεψη για το κλίμα στο Παρίσι, πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνούμε με την πρόταση αυτή. Αλλά όπως είπε και ο σοσιαλιστής συνάδελφος, εγώ και εγώ θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια Έχω πιστοσύνη βέβαια σε την πραγματεύσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω να μην ε, κρύβεται κάποιος διάβολος στις λεπτομέρειες ε, που θα μας ε, δημιουργήσει πρόβλημα στην πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήθελα να πάρω το λόγο γιατί θυμάμαι την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε. Η πρόταση σύνδεσης μεταξύ των δύο συστημάτων ε, εμπορίας δικαιωμάτων αερίων θερμοκηπίου. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη έκθεση είναι ένα καλό βήμα προς τα εμπρός, ώστε να εξασφαλίσουμε ώστε κάθε χώρα και κάθε κλάδος ε, που συμβάλλει στην μόλυνση ε, να μπορέσει να ε, συνεισφέρει και στη μείωση της ε, μόλυνσης. Συγκρίνοντας τα δύο συστήματα βλέπουμε ότι η δομή είναι παρόμοια. Ακολουθούμε τις ίδιες αρχές και μπορούμε επίσης να πούμε Τα συστήματα μας πάνε από το 2013 μέχρι τις 2020 όσον αφορά ε, τη μείωση ώστε, τη μείωση των εκπομπών αερίων, ώστε ε, ε διεθνώς κάθε χρόνο να μειώνονται οι εκπομπές ε, αερίων θερμοκηπίου. Θα ήθελα να τονίσω το εξής. κυρίως αυτό που είπε ο συνάδελφος Παρνιό ε, και να συμφωνήσω μαζί του, θα θέλαμε περισσότερη διαφάνεια. Θα θέλαμε να ξέρουμε τους τομείς που καλύπτονται, όπως επίσης και πληροφορίες σε σχέση με άλλες ενδεχόμενες συμφωνίες. Ευχαριστώ πολύ. Και τι δυνατότητα έχουμε σύνδεσης με άλλα συστήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες ε, στον ε, ε, εισηγητή, όπως επίσης και σε όλους όσους μας υποστηρίζουν στην πρότασή μας. Πράγματι, θεωρούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και έγκαιρο, επίκαιρο βήμα ε, η σύνδεση του συστήματός μας με της Ελβετίας, δύο συστήματα εκπομπών ε, ε, διοξιδίου του άνθρακα και για να μπορέσουμε να διευρύνουμε τις αγορές και να μπορέσουμε να επιτύχουμε από κοινού τους μακροπρόθεσμους στόχους μας. Τώρα υλοποιείται για πρώτη φορά, γιατί η Ελβετία που έχει ένα πολύ παρόμοιο σύστημα σε σχέση με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πρόθυμη να το κάνει και να απαντήσω στο ερώτημα που μόλις άκουσα για τους κλάδους. Ε, οι ίδιοι κλάδοι καλύπτονται και από την ελβετική πλευρά. Θέλουμε να καλύψουμε και την αεροπορία. Αυτό κάνουμε τώρα στις διαπραγματεύσεις μας με τους Ελβετούς. Οι ε, ίδιοι κλάδοι λοιπόν, ε, συν την αεροπορία που προσπαθούμε να επιτύχουμε την περασμένη εβδομάδα, μπορεί και να το είδατε στο τύπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επέγραψε τη συμφωνία που είναι το πρώτο διαδικαστικό βήμα που πρέπει να κάνει. Ο πρόεδρος Γιούνκερ και, και η κυρία Λάρτσατ ε, από την ελβετική πλευρά. Πράγματι αυτό είναι μια πολύ ευχάριστη ε, εξέλιξη μία μέρα μετά που το Συμβούλιο ενέκρινε την προσωρινή ε, συμφωνία για την ε, συνέχιση του συστήματος ε, εμπορίας εκπομπών αερίων. Το ETS λοιπόν είναι το μεγαλύτερο σύστημα εμπορίας αερίων στον κόσμο και δείχνει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί και με άλλους εταίρους ε, που επίσης παίρνουν εξίσου σοβαρά ε, τις, ε, τους στόχους αυτούς και θέλουμε επίσης να τιμολογήσουμε και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τον άνθρακα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να επανέλθω τώρα στη σχέση μας με την Ελβετία, όπως είπα, έχει ήδη υπογραφεί η συμφωνία. Ελπίζουμε και εσείς να την εγκρίνετε και την εφαρμογή της. Βεβαίως, το Συμβούλιο ετοιμάζονται για την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Υπάρχει λοιπόν ε, το θέμα της έγκρισης των συμπερασμάτων. Όταν θα γίνει αυτό θα μπούμε σε προπαρασκευαστικές συζητήσεις με την Ελβετία για να είμαστε έτοιμοι για τη σύνδεση των συστημάτων. Η ίδια η συμφωνία Αφού εγκριθεί η πρόταση για σύναψη της συμφωνίας, ε, δεν θα αρχίσει να ισχύει πάρα πολύ σύντομα. Θα πρέπει να ε, εργαστούμε προς την ετοιμότητα όσον αφορά τα μέσα που χρειαζόμαστε και τα μέσα που θα μας βοηθήσουν να ευθυγραμμιστούμε, να συνεργαστούμε με την ελβετική πλευρά, ε, δηλαδή πώς μπορούν πράγματι να συνδεθούν τα συστήματα ε, και από πλευράς μας και από την Ελβετία. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει διασφάλιση ότι όλα αυτά τα οποία υποσχέθηκαν οι Ελβετοί να κάνουν, δηλαδή να συμπεριληφθεί στο δικό τους ETS η αεροπορία ότι θα το έχουν κάνει, θα πρέπει να το ελέγξουμε αυτό και μετά πρέπει να γίνει και ο έλεγχος συμμόρφωσης και τότε θα είμαστε σε θέση να ε, υποβάλουμε το ε, μέσο μας προς ε, έγκριση προς επικύρωση μάλλον. Όπως είπατε και εσείς, είναι πάρα πολύ μεγάλη πολιτική σημασία αυτού του, αυτής της συμφωνίας. Σε μία χρονική στιγμή, όπως είπατε και εσείς, που η αγορά ε, άνθρακα είναι πάρα πολύ δυναμική, υπάρχουν ε, πολύ μεγάλες εξελίξεις σε όλο τον κόσμο, βλέπετε την Κίνα ε, και το ακούσαμε και στη Βόνη αυτή στο πλαίσιο της COP23 στα τελευταία στάδια του εθνικού της ETS βρίσκεται και όπως ξέρετε συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με την Κίνα προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο αλλά υπάρχουν και άλλες εξελίξεις όπως στον Καναδά για παράδειγμα ή στις Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι λοιπόν ε, ένα πολύ δυναμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να στείλουμε και αυτό το μήνυμα επιπλέον τη σύνδεση με το ελβετικό ETS. Ε αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό για να προετοιμάσουμε το έδαφος για μια παγκόσμια αγορά είναι να δουλέψουμε και με τρίτες χώρες που θέλουν να το αναπτύξουν αυτό και σε εγχώριο επίπεδο και αυτό θα είναι αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει. Κάποιες χώρες είναι αρκετά προχωρημένες, είναι στο στάδιο της εφαρμογής, άλλες είναι στο στάδιο της ανάπτυξης μόνο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε πολύ στενά μαζί τους για να εξασφαλίσουμε ότι θα αναπτύξουν ισχυρά και ανθεκτικά συστήματα ε, και μετά να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να ε, εξετάσουμε τη σύνδεση μαζί τους. Δεν θα γίνει αύριο αυτό, ίσως μεθαύριο. Και ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι σημειώνω το αίτημά σας για διαφάνεια, για περισσότερη διαφάνεια. Θα το έχουμε υπόψη μας για τις μελλοντικές μας συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπέλετ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώς να πω ότι συμφωνώ με όλα και ιδίως τον κύριο Παρνιό, κυρία Ντάλη, την κυρία Κονέτσνα, Είναι μεγάλο βήμα πρόοδο Και έχει δίκιο ο κύριος Παρνιό να βρω ότι δεν υπάρχει διαφάνεια και ότι θα μπορούσε να υπάρχει περισσότερη ενημέρωση, να έρχεται πιο γρήγορα αυτή η ενημέρωση. Ε, ελπίζω ότι αυτό να είναι ένα συμπέρασμα το οποίο να αντιληθεί από όλα τα θεσμικά όργανα και το οποίο και η κυρία Κονίζα ότι αυτό είναι ένα μικρό βήμα προς τον υπάρξει ένα παγκόσμιο τελικά σύστημα. Τα συζητήσαμε στη γόνη και με τους Κινέζους. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπουν στο παιχνίδι και οι Κινέζοι. Άρα ελπίζουμε ότι με αυτό το βήματάκι θα αλλάξουμε ρότα και μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την αίσια κατάλληλη τη διαδρομή. Ε, ευχαριστούμε, μπράβο, καλά τα πήγατε, μπράβο, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα, αν έχετε κάποιε τροπολογίε, βιαστείτε. Έξι ώρα. Απόψε εκπνέει η προθεσμία. Και θα ψηφίσουμε αύριο. Uh, Έχουμε το, το, άλλο θέμα. Όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, την ε, το του Κοινοβουλίου, το πολιτές πλαίσιο για μετά το 2020, η κυρία Γιατενμάκη είναι η, εισηγήτρια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι. Rahoituskausi päättyy siis 2020 mennessä. Ja Είπαμε ότι το Κοινοβούλιο θα τοποθετηθεί σε σχέση με την ε, ε, έκθεση αυτή που θα συντάξει η Επιτροπή Προπολογισμών, οπότε και η Επιτροπή μας αυτή θα εξηγήσει το ποιες είναι οι προτεραιότητες, θα προβεί στη προσχετική πρόταση ε, και αυτό το πολιτές δημιουργικό πλαίσιο, το MFF, είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντοτε ήταν και τώρα έχουμε περισσότερο, μια που <coughs> έχουμε συγγνώμη το Brexit, το οποίο είναι μια δαμόκλειος σπάθη στον προπολογισμό και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε, σε τι σχέση θα καταλήξουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο, αν υπάρχει καμία σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο Πάντως στην Επιτροπή μας αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τα ζητήματα που μας αφορούν. Οπότε έχουμε και υποχρέωση να τοποθετούμε για το MFF. Πάντως υπάρχει κάποια έκπληξη, προσδοκούσαμε περιμέναμε τέλος πάντων αυτές τις προτάσεις της Επιτροπής και κοιτώντας προς το μέλλον θα πρέπει να τοποθετηθούμε να πούμε τι θέλουμε να πετύχει αυτό το πολιετές πλαίσιο. Τι θέλει η Επιτροπή μας. Τι περιμένει από αυτό το MFF. Δεν να λάβουμε υπόψη τι με τα προηγούμενα δημοσιονομικά πλαίσια, τι έπιασε τόπο, τι επιδεχόταν βελτίωση κλπ. Διότι θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και σε μερικέ περιπτώσει θα πρέπει να γίνεται όπω θα περιμέναμε. Άρα, πιάσουν από τα λεφτά, θα πρέπει ό,τι κάνουμε να κατευθύνεται προ την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Ε, είπαμε να έχουμε μια οικονομία που να μην χρησιμοποιεί τον άνθρακα, θα πρέπει να έχουμε καταναλώση ενέργεια που να είναι βιώσιμη και με τον προπολογισμό μα θα πρέπει να προωθήσουμε κάποιε λύσει φιλικέ στο περιβάλλον, να βοηθούμε τη δημοσία υγεία και όλα τα σχετικά. και την βιοπικιλότητα να βοηθούμε. Είναι σαφές ότι αυτό το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο πρόκειται να αμφισβητηθεί μια που και το τρέχον, το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο δεν μας επέτρεψε να κάνουμε όλα όσα θέλαμε να καλύψουμε αυτά που φιλοδοξούσαμε και έχουμε τις σχετικές υποσχέσεις ε, των Παρισίων είπαμε ότι με το 2020 θέλουμε να μειώσουμε τι εκπομπέ που δεν θα το καταφέρουμε. Έχουμε δεδομένε προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να δούμε εάν θα μπορούσαμε τελικά να πετύχουμε κάποιου στόχου για το περιβάλλον. Σίγουρα θα πρέπει βέβαια και οι στόχοι μας να τίθενται με προσοχή, να υπάρχει διαφάνεια. Νομίζω ότι αν θέλουμε μπορούμε να πετύχουμε αυτά προς το παρόν και περιμένω να ακούσω τις ε, απόψεις σας. Η Πρόεδρος. Ε. Ευχαριστούμε. Θα δώσω τώρα το λόγο στους ε, με πρώτον τον κύριο Κοβάτσεφ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τεμάκη. Είναι πολύ καλή αφετηρία το έγγραφό της για τη συζήτηση για το ΠΔΠ μετά από τις σημαντικές εξελίξεις έχουμε ε, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στη συζήτηση που έχει ξεκινήσει που είναι ο προπολογισμό μετά το 2020 γιατί δεν μπορούμε να φέρουμε σε πέρα σε όλες τις προτεραιότητες μας αν δεν έχουμε ένα επαρκές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά την ε, ολοκλήρωση της Συμφωνίας ε, των Παρισίων η καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής έχει προσλάβει πολύ μεγάλη σημασία, πιο πολύ από ποτέ. Πρέπει να παραμείνουμε σε πρώτη, στην πρώτη γραμμή και θα πρέπει με τον προπολογισμό μας να στηρίξουμε την ταχεία εφαρμογή τη Συμφωνία των Παρισίων, να προωθήσουμε τη μετάβαση καθαρή ενέργεια, την απαλλαγή από άνθρακα τη οικονομία μα, να προωθήσουμε την κυκλική οικονομία και να υπογραμμίσουμε ότι το πολιετέ το επόμενο θα πρέπει να συνεισφέρει και στην ε, επίτευξη των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Ένωση για τους, βιώσιμους, ε, μάλλον για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Το μερίδιο του προπολογισμού που θα διατεθεί σε θέματα συνοχής δεν θα πρέπει να μειωθεί μετά το 2020. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο Ταμείο Συνοχής ε, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή ανάπτυξη και άλλα διαρθωτικά ταμεία είναι σημαντικά για να μειώσουν τι ανισότητες μεταξύ περιφερειών και να βελτιώσει το περιβάλλον στις λιγότερο ανεπτυγμένες ε, περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωση. Βέβαια, αυτό πρέπει να συμβαδίζει και με τη διερεύνηση νέων ε, τρόπων αξιοποίηση των εργαλείων που βασίζονται στην αγορά για την επιτέξη των στόχων μας τέλος. Δεν μπορεί κανένα κράτος μέλος από μόνο του να αντιμετωπίσει τις συνολικέ προκλήσεις. Γι' αυτό και πιστεύω ότι το πολιτέ θα πρέπει στο μέλλον να αντικατοπτρίζει την ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να στηρίζει τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν τάσεις οι οποίες ε, θα υποβαθμίσουν ή θα απονομεύσουν την ε, συνοχή. Έχουμε τι μεταδοτικέ ε, νόσου. Έχουμε επιδημίες, έχουμε παχυσαρκία, ε, την αντοχή στα μικρόβια και στα αντιβιωτικά, επιδημίες. Όλα αυτά απαιτούν να εξασφαλίσουμε την ισότιμη πρόσβαση όλων σε, σε υπηρεσίες υγείας και αυτό βέβαια και μετά το 2020. Περιμένω να συνεργαστώ ε, με τους συζητητές, τους και σας ευχαριστώ. Uh, ναι, και εμείς προσβλέπουμε στην μεταξύ μας εργασία. Η κυρία Ντάλη δεν είναι ο σκιός εδώ, αλλά είναι η κυρία Ντάλη. Είναι πολύ σημαντικό θέμα, ε? βεβαίως, κυρία Πρόεδρε. Ναι, και καταρχάς να ξεκινήσω από τη θέση της, του σκιώδους του κυρίου Καπούτο που δεν είναι εδώ. Και μετά θα σας πω τις δικές μου απόψεις, αλλά καταρχάς θα σας αναφέρω τις απόψεις του κυρίου Καπούτο, ο οποίος πρώτα απ' όλα θέλει να ευχαριστήσει την κυρία Τεμάκη για ε, τη θετική της προσέγγιση σε αυτή τη γνωμοδότηση. Γίνεται αναφορά στις προτεραιότητες της Ένωσης και στις εξωτερικές δεσμεύσεις και στην ανάγκη συνέχισης των πολιτικών βιωσιμότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Οι τροπολογίες που θα καταθέσει ο κ. Καπούτο για τα στήματα αυτά θα έχουν ως στόχο ε, κάποιες διευκρινήσεις, κάποια βήματα. Πρώτον, θεωρεί ο κ. Καπούτο ότι δεν γίνεται αναφορά στην κυκλική οικονομία ούτε στα καινοτόμα σχέδια στον τομέα αυτό. Μερικά έχουν να κάνουν και με το Horizon 2020 και με το LIFE. Επίσης θεωρεί ότι το LIFE θα πρέπει να έχει την απαραίτητη υποστήριξη για να βελτιωθεί η εφαρμογή του ιδίω σε ολοκληρωμένα σχέδια. Η Ευρώπη είναι ηγέτης στον κόσμο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ε, και στις περιβαλλοντικές πολιτικές πρέπει να συντονίζουν τα κράτη-μέλη τις πολιτικές τους. Γι' αυτό, παρά το Brexit, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα βήμα προς τα πίσω σε τεφά τις πολιτικές αυτή Τέλος. Ένα πολύ στενά συνδεδεμένο θέμα είναι το θέμα των ιδίων πόρων. Πρέπει να βρούμε πρόσθετους πόρους για να μην κάνουμε ένα βήμα πίσω σε τεφά τις μελλοντικές πολιτικές και προκλήσεις για τις οποίες έχουμε τη χαράξει το δρόμο και τώρα αυτό που χρειάζεται είναι να δείξουμε το απαραίτητο στένος για να προχωρήσουμε. Δεν μιλάμε μόνο για τι εσωτερικέ, αλλά και τι εξωτερικέ δράσει τη Ένωση. Θα πρέπει να δοθούν κονδύλια και στι αναπτυσσόμενε χώρε. για να μην μείνουν σε παλιές τεχνολογίες και να μην ε, ακολουθήσουν έτσι την εσφαλμένη προσέγγιση των ε, κρατών μελών. Είχαμε επίσης ε, φυσικές καταστροφές και ιδίως στην Ιταλία, την πατρίδα του κυρίου Καπούτο, αλλά και σε, με τους σεισμούς, αλλά και σε άλλες χώρες τη Ένωση, που δείχνει ότι Υπάρχει αυτό το σύστημα συντονισμού που λειτουργεί, αλλά πρέπει να βελτιθεί περισσότερο. Και βέβαια, πολιετές ε, διάρκεια του πολιτού. είναι ένα θέμα που πρέπει να μα απασχολεί. Αν έχουμε πάνω από πέντε χρόνια και υπάρχει και η δυνατότητα αναθεώρησης, θα βοηθήσει αυτό σχέδια που έχουν ευρύτερο ορίζοντα, όπως τα σχετικά με το κλίμα. Τώρα, αν μου επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω μαλτέζικα για να σας πω τα δικά μου σχόλια. Καταρχάς, θέλω να πω ότι συμφωνώ με την εισηγήτρια που στην πρώτη παράγραφο ιδίω λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διαρθρώσει κατά τέτοιο τρόπο το επόμενο ΠΔΠ που να αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες της Ένωσης. Και ιδίως ό,τι αφορά την ανάγκη ο ρόλος της Ένωσης ότι αυτή την κλιματική αλλαγή να παραμείνει εξίσου σημαντικός και κεντρικός. Θέλω επίσης να ψήσω την προσοχή σας στο πράσινο ταμείο χρηματοδότης και ποιος είναι ο ρόλος μας σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση αυτού του ταμείου. Αυτό το ταμείο ίσως είναι ο πιο πρόσφατος ε, ε, παράγοντας σε αυτή την αρχιτεκτονική χρηματοδότηση ε, του κλίματος και θα είναι πλήρως επιχειρησιακό σύντομα. Έπρεπε να είναι το 2015. Και ο στόχος είναι να διοχετεύσει πόρους στις αναπτυσσόμενες χώρες και να δράσει ως καταλήτης για την προσέλκυση ιδιωτική χρηματοδότησης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Βέβαια, βλέπουμε δυστυχώς ότι ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Συμφωνία των Παρισίων. Σε αυτό το πράσο ταμείο για το κλίμα υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις που δεν θα υλοποιηθούν. Μιλάμε για δύο δις δολάρια. Μπορεί να είναι και πολλά ε, αν τα δει κανεί ε, σφαιρικά τα πράγματα, όμως έχει πολλές ε, επιπτώσεις στο μέλλον που δεν μπορούμε να τις συνειδητοποιήσουμε τώρα η τρύπα αυτή των δύο δις. Το θέμα είναι να βρούμε καθαρή ενέργεια και με περαιτέρω χρηματοδότηση να βοηθήσουμε αγορές που θα δράσουν ως καταλήτη την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, για τη μεγάλο μέρος των επενδύσεων για το πράσινο ταμείο το κλίμα έχει κάποια επιστροφή οικονομική, δηλαδή τα χρήματα που δίνουν σε αυτό το ταμείο μπορούν να βοηθήσουν για την ε, δημιουργία περισσότερων του ενός προγραμμάτων και σχεδίων. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνω έκκληση. Όταν κοιτάμε προς το μέλλον, να φροντίζουμε η δημοσιονομική πολιτική της Ένωσης τα επόμενα 7 χρόνια να είναι και αυτή επαρκής και προσαρμοσμένη στο επόμενο πολυετές που ελπίζουμε να διαρκέσει 7 χρόνια. Ευχαριστώ. Thank you very much. Very Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιδέα. Now, uh, Konechna, Κυρία Κονέτσινα, θέλετε να πάρετε το λόγο? Όχι. Καλώς. Ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Βουριό. Yes, you have the floor. Um, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ στην εισηγήτρια για την γνωμοδότηση αυτή και για την ανταλλαγή απόψεων. Πράγματι, όπως είπε και η κυρία Γιατενμάκη, είναι Μία πολύ σημαντική στιγμή για τον προβληματισμό ως προς το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε τη διαδικασία με τη Λευκή Βίβλιο το Μάρτιο αλλά και με το έγγραφο προβληματισμού τον Ιούνιο για τα οικονομικά της Ένωσης στο μέλλον. Η, Ευρωπαϊ... η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω της έκθεσης ε, ε, ε, ε πρωτοβουλίας μεταξύ ε, ε, από τον κύριο Όλμπριχτ ε, θα είναι πάρα πολύ σημαντική εν ώψη της προετοιμασίας του πλαισίου αυτού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τα, τις προτάσεις της το Μάιο του 2018. Όπως γνωρίζετε, οι προτάσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ουσιαστικά συμπεριλαμβάνουν ένα ευρύτερο πλαίσιο όσον αφορά και, τον, και το ε, πλαίσιο το χρηματοοικονομικό αλλά και ε, τα μέσα πολιτικών ε, είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά της Επιτροπής σας για την αξιολόγηση του LIFE για παράδειγμα ε, ή προγραμμάτων ε, για το κλίμα και για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είδατε, επειδή έχουμε ήδη δημοσιεύσει κάποιες ενδιάμεσες ε, αξιολογήσεις των προγραμμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, χρησιμοποιεί και ε, προβληματίζεται βάσει αυτών των εγγράφων. Περιμένουμε λοιπόν εναγωνίω την ε, συζήτηση και τη συμμετοχή σας. Συζήτηση με εσά και τη συμμετοχή σας. Κυρία Γιατενμάκη. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις πάρα πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις και σχόλιά τους. Θα τις λάβω υπόψη όπως και τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 5 Δεκεμβρίου, 21 Ιανουαρίου ψηφίζουμε στην ΕΝΒΗ. Και πάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι οι γλυκαντικές ουσίες στα αρτοσκευάσματα. Λοιπόν, εξέταση πρότασης ψηφίσματος ε, για την αντίρρηση αυτή. Η κυρία Γκροστέτ το έχει αναλάβει, αλλά νομίζω η κυρία Γιούσο την ε, αντικαθιστά. Ή όχι. Όχι. Α, ο κύριος Μπέλετ. Κύριε Μπέλετ, τώρα έχετε και τις γλυκαντικές ουσίες να μας παρουσιάσετε. Έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε την αντίρρησή σας. Ναι, βεβαίω. προτεραιότητα έπρεπε να δώσω σε έναν από τους αντιπροέδρους τη Επιτροπής μου. Εκ μέρου λοιπόν της κυρίας ε, Γκροστέτο, όσον αφορά τη χρήση γλυκαντικών ουσιών στα αρτοσκευάσματα. Να σα πω μερικά στοιχεία. Καταρχάς, να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να αξιολογήσει τις ε, συνέπειες της ανάκλησης της οδηγίας ε, για ε, τις γλυκαντικές ουσίες στα τρόφιμα, οπότε όλες αυτές οι γλυκαντικές ουσίες για τις οποίες μιλούμε θα παραμείνουν, θα εξακολουθεί να ισχύει η άδειά τους για τη χρήση στις μαρμελάδες, σε κάποια ποτά, αλλά θα απαγορεύονται στάρτος αρτοσκευάσματα για τα οποία γίνεται λόγο σήμερα. Αυτά τα αρτοσκευάσματα, ε, τα οποία έχουν σκοπό βέβαια να καταναλώνονται ως διατροφικά προϊόντα ε, από τον άνθρωπο και ε, κατά τη γνώμη μας από απόψεις δημόσιας υγείας δεν έχει κανένα νόημα. Προτείνουμε Ε, αυτό που προτείνουμε το προτείνουμε γιατί δεν υπάρχει μεταβατική περίοδος που να προτείνεται και αυτό θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπάρχει η μεταβατική περίοδος θα απειλήσει τη διαθεσιμότητα προγραμμάτων αυτών όπως ε, τα κέικ, τα κούκκι, τα μπισκότα δηλαδή ε, και τις μπάρες που έχουν, δεν έχουν καθόλου ζάχαρη και είναι ένα πρόβλημα για όλους όσους χρειάζονται μια δίαιτα χαμηλών λιπαρών χωρίς ζάχαρη όσους έχουν διαβήτη. Οι γλυκαντικές ουσίες που χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα είναι οι μόνες που επιτρέπονται ε, ως εναλλακτική λύση σε ε, υψηλή περιεκτικότητα ζάχαρη. Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας η νομοθεσία να προβλέπει μία εύλογη περίοδο μεταβατική ε, και όχι κατευθείαν απαγόρευση. Δύο χρόνια μεταβατική περίοδο, τουλάχιστον ώστε αυτέ οι γλυκαντικέ ουσίε να μπορέσουν ε, να αν ε, να δομηθούν και να μπορέσουν να ξαναδιατηθούν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις διατροφικές ανάγκες κάποιων πολιτών. Δεν θα πω τώρα σε πολλές λεπτομέρειες ε, ε, ως προς το επιχείρημά μου, αλλά μου φαίνεται ότι είναι λογικό ε, γιατί έχει πάρα πολλές συνέπειες για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον, στους, στους τομείς τους σχετικούς. Προτείνουμε λοιπόν αυτή την αντίρρηση βάσει αυτών των λόγων εκ μέρου της ε, εισηγήτρια της Φρονσουάς Γκροστέτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι, η κυρία Γιούσο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο για να συμφωνήσω με τα όσα έχει προτείνει η κυρία Γκροστέτ και όπως τα προτείνει είναι θέμα δημοσίας υγείας. Είναι ασφαλείς αυτές οι ουσίες. Τόσα χρόνια είναι στην αγορά. Έχουν περάσει από έγκριση για τη χρήση τους σε διάφορα είδη διατροφής. Και είπαμε ότι θέλουμε τώρα να αλλάξει αυτή η νομοθεσία για διάφορες κατηγορίες των διατροφής, αλλά σε αυτή την περίπτωση η Κομισιόν πρόκειται από τους διαβητικούς να στερήσει αυτά τα προϊόντα. Και επίσης, όπως είπε και ο κύριος Μπέλετ, θα δημιουργήσει πρόβλημα και σε πολλές έψιλων. Ε. επομένως υπάρχουν πολλά επιχειρήματα για να συμφωνήσουμε με την πρόταση. Άλλος θέλει το λόγο, λέει πρόεδρος, όχι, επομένως, κύριε Γιούλη, κύριε, έχει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. να αναφερθώ στις προϋποθέσεις έγκρισης πρόσθετων ουσιών. Το είπαμε και προηγουμένως για τα φωσφορούχα. Οι προϋποθέσεις προβλέπονται από την οικία νομοθεσία. Δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία. Θα πρέπει να υπάρχει ανάγκη δημιουργημένη επιστημονικά. Θα πρέπει να είναι παραπλανητικό για τον καταναλωτή, θα πρέπει να τον ωφελεί. Όσον αφορά την έγκριση της χρήσεως των ελκαντικών ουσιών θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον μία από τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως ορίζονται από την σχετική νομοθεσία για τις πρόσθετες ουσίες ή στα τρόφιμα. Οπότε αυτές οι προϋποθέσεις είναι την, να, να αντικαταστήσουν την ζάχαρη για κάποια ειδικά οι διατροφείς που δεν πρέπει να έχουν ζάχαρη ή θα πρέπει να παρατηρούν την διάρκεια ζωής του προϊόντος, να απευθύνεται σε συγκεκριμένους ε, χαριστες όπως ορίζει ε, η οδηγία Αυτό είναι το κείμενο νομικό πλαίσιο και έχουμε τις σχετικές τροποποίησεις γιατί στο παρελθόν ε, αυτού του είδους τα προϊόντα που είχαν χρήσει οι ειδικοί είχαν εγκριθεί με την οδηγία 94-35 γιατί αφορούσαν ε, συγκεκριμένους αποδέκτες συγκεκριμένους χρήστες όπως ορίζει 89-38 και είπαμε ότι οι διαβητικοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους ε, ε τρόφιμα όπως ορίζει η οδηγία του 89 τροποποιήθηκε η οδηγία αυτή και είπαμε ότι θα μπορούσαν να θεσπιστούν συγκεκριμένες διατάξεις για συγκεκριμένες διατροφές για τους διαβητικούς. Το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε κάποια μελέτη για τους διαβητικούς και τα σχετικά τρόφιμα λέγοντας ότι δεν υπάρχει ψημιλική βάση ούτως ώστε να τεθούν προϋποθέσεις για αυτά τα τρόφιμα. Οπότε και προχώρησε στη σχετική νομοθεσία χωρίς τέτοιες προϋποθέσεις. Έχουμε την οδηγία 1939 που δεν ισχύει πλέον στα πλαίσια της ενίας αγοράς. Αφορά τα τρόφιμα ειδική χρήσης και αφορά και τα τρόφιμα για διαβητικούς. και ο κανονισμός 13 του Συμβουλίου Κοινοβουλίου καταργήθηκε. Εδώ είναι τώρα το πιο σημαντικό. Γιατί αυτή η αλλαγή στην νομοθεσία προκάλεσε όλα όσα έγιναν. Ξεκίνησε αυτό το 2013 με τον 609 του 13. Τόσα ισχύει το 2016. και όλοι οι εμπλεκόμενοι και η βιομηχανία ενημερώθηκε. Οπότε, αφού πια έχουν απαλληφθεί από αυτή την νομοθεσία τα, αυτά τα ειδικά τρόφιμα για τους διαβητικούς, δεν υπάρχει δικαιολόγηση ούτε λόγος να υπάρχει αυτή η ομάδα προϊόντων που συζητούμε τώρα. και ούτε αυτή η ρύθμιση για αυτές τις γλυκαντικές ουσίες. Από το 2013 επομένως αυτή η έννοια δεν δικαιολογείται να καλύπτεται την νομοθεσία. Ούτε όμως και να τίθεται σε εμπορία τέτοιο προϊόν. Επομένως, θα πρέπει να τροποποιηθεί αυτός ο κανονισμός όσον αφορά αυτές τις γλυκαντικές ουσίες για αυτά τα προϊόντα και τα αρτοσκευάσματα. Εμείς σεβαστήκαμε την αρχή της αναλογικότητας και προτείνουμε μεταβατική περίοδο για την βιομηχανία. Επομένως, αυτό το σχέδιο κανονισμού συνάδει με όσα προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο για τα γλυκαντικές ουσίες. Και τα όσα η επιστήμη προβλέπει και περιέχονται στον Οργανισμό 609 του 13. Αυτή είναι η επιστημονική αξιολόγηση. Ότι οι διαβητικοί θα πρέπει να ακολουθούν μια υγιεινή διατροφή, αλλά να διατρέφονται με φυσιολογικά τρόφιμα. διαβήτης ε, Β, ε, υπάρχει σαρκία και αυτά καλύπτονται από κάποια τρόφιμα που έχουν φυσικές ίνες, αλλά αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τον διαβήτη. Και επίση κάποια προϊόντα έχουν ε, υδατάνθρακες και ακριβώς μιλούμε για αυτά τα, αυτά τα αρτοσκευάσματα για τα οποία θα πρέπει να σας πω ότι αυτός ο κανονισμός δεν αποτελεί φραγμό στην καινοτομία. Όπως είπαμε, αυτή η ρύθμιση ξεκίνησε το 2013. η καινοτομία δεν σημαίνει μόνο να προσθέτονται τα αγγλικαντικά. Είναι και το να ε, θέτει κανείς σε εμπορία αρτοσκευάσματα που να έχουν λιγότερη ζάχαρη, ε, υδρογονωμένα λίπη κλπ. βιομηχανία, όπως είπαμε, είχαν αρκετό χρόνο μετά τη θέσπιση του κανονισμού του 2013. Το 2016 ετέθησε ισχύ αυτός ο κανονισμός και αυτή η μεταβλητική περίοδος δόθηκε και ρητός προβλέφθηκε από τον κανονισμό. Σε αυτή την περίοδο είπαμε ότι αυτά τα αρτοσκευάσματα για ειδικού χρήστες νομίμως τέθη εμπορία πριν τον κανονισμό. Μπορεί να συνεχίσουν να πολλούν και να θέτουν εμπορία αυτά τα προϊόντα μέχρι να εξελιχθούν τα αποθέματα και εμείς πάντως πιστεύουμε ότι αυτό το σχέδιο κανονισμού είναι σύντονο προς την αρχή της αναλογικότητας και αυτό θα γίνει όταν εφαρμοστούν οι προϋποθέσεις με ομοιογενή τρόπο. Σύμφωνα με τις νόμιμες πρακτικές με την του λειτουργία της μενίας ε, αγοράς και έτσι να υπάρχει ασφαλή δικαίου για όλους τους εμπλεκομένους να προστατεύονται και τα συμφέροντα του καταναλωτού. Και επίσης δόθηκε αρκετός χρόνος για προσαρμογή στη νέα κατάσταση μετά την τροποποίηση του 13. Οπότε είναι ενδεδειγμένη αυτή η μεταβατική περίοδος και καλύπτει και τα προϊόντα τα οποία νομίζω, έχουν τεθεί σε εμπορία. Ε, ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Σαλντεμόσε. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που άργησα λίγο και δεν άκουσα το πρώτο κομμάτι της συζήτησης γιατί είχα μια ομάδα επισκεπτών. Θα ήθελα να πω ότι η ομάδα μου δεν στηρίζει αυτή την αντίρρηση δεν στηρίζουμε την αντίρρηση, διότι θεωρούμε πως οι επιχειρήσεις είχαν τον απαιτούμενο χρόνο να προσαρμοστούν στην νομοθεσία αυτή. Θεωρούμε επίσης ότι πρόκειται για μια φυσική απόρρεια της νομοθεσίας, η οποία εγκρίθηκε το 2013. Είναι λογικό και επόμενο να μην περιλαμβάνονται αυτές οι γλυκαντικές ουσίες στα, αυτά, στα ειδικά αυτά τα σκευάσματα. Θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις πλέον γνωρίζουν την νομοθεσία και είχαν δυνατότητες να μπορούν να παρασκευάζουν άλλα ε, τέτοια τρόφιμα με άλλους τρόπους. Δεν μιλήσαμε επίσης πολύ για τους διαβητικούς και τις ε, ενώσεις διαβητικών. Δεν έλαβα κάποια αντίρρηση από τις ε, ενώσεις των διαβητικών, άρα θεωρώ ότι μπορεί κανείς ε, να τρέφεται υγιεινός χωρίς να χρειάζεται αυτή η πρόταση. Δεν ήθελα να ξαναρχίσει η συζήτηση, δεν ήταν αυτή η προθεσμή μου, αλλά το κάνατε εσεί, κυρία Σαλντεμόζη. Ουσιαστικά, όποιο θέλει λοιπόν το λόγο μπορεί να τον πάρει. Κυρία Ζόμερ, πρώτη. Κυρία Ζόμερ, δεν είπατε ότι θέλετε το λόγο. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά ε, τη νομική κατάσταση του θέματος, ε, γνωρίζω τα πράγματα και καλά λέει η Κομισιόν ότι ε, υπάρχουν αυτά τα τεχνικά επιχειρήματα που λένε ότι αυτά τα κλικαντικά ότι αυτά ε, θα πρέπει πλέον να χρησιμοποιούνται. Δεν μιλάμε όμως μόνο για τους διαβητικούς, αλλά και για παχύσαρκους και όταν αυτά τα αρτοσκευάσματα ε, δεν ε, μπορούν πλέον να καταναλωθούν από αυτά τα άτομα είναι κρίμα γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι τους βοηθούν ε, αυτά τα προϊόντα και τα χρησιμοποιούσαν. Όταν λέει κανείς τώρα στους διαβητικούς ότι πρέπει να τρέφονται κανονικά και δεν χρειάζονται ειδικά προϊόντα, όμως ε, για το τους παχύσαρκους ε, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ε, δεν πρέπει να τρώτε καθόλου γλυκά ή ψωμιά ή οτιδήποτε αμυλούχο. Γιατί μπορεί να υπάρχουν συνταγές που περιλαμβάνουν λιγότερο αλάτι, λιγότερη ζάχαρη, λιγότερη ε, δεν ξέρω εγώ τι υδατάνθρακες, ε, αλλά αν τα αφαιρέσουμε όλα δεν τελικά πάνε τα προϊόντα, δεν θα μπορούμε να φτιάξουμε τίποτα ε, ως αρτοσκεύασμα πλέον που να μπορεί να διατίθεται. Για τους παχύσαρκους ε, θα μπορούσε να είναι βοηθητικό πιστεύω να παραμείνουν στην αγορά τέτοιου είδους προϊόντα πέραν των ε, διαβητικών, γιατί ξέρω την, ε, το νομικό καθεστώς ε, πολύ καλό, νομίζω ότι είναι λογικό αυτό που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τεχνικής πλευράς, όμως ναι, δεν, δεν μπορούμε να το δούμε μόνο έτσι το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριο Μπέλετ. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρου τη κυρία Γκροστέτ. δεν έχουμε να προσθέσουμε πολλά στα όσα είπα η κυρία Ζόμερ και άλλοι υπέρ της ε, αντίρρησης δηλαδή. Δεν αμφισβητούμε αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν αμφισβητούμε τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βέβαια. Μιλάμε για τα συμφέροντα των καταναλωτών. Εκεί δεν πολύ συμφωνούμε. Εντάξει, η νομική, η ασφάλεια δικαίου και τα λοιπά, ναι, φυσικά. Καλό επιχείρημα και το ενστερνιζόμαστε. Όπως είπε και η κυρία Ζόμερ όμως, αυτό σημαίνει τελικά βραχυπρόθεσμα, αυτά τα αρτοσκευάσματα δεν θα είναι διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή αγορά. Και μιλάμε για ευρωπαίους καταναλωτές. Όχι διαβητικούς μόνο, όπως είπε και η κυρία Ζωμέρα, ε, αλλά και παχύσαρκους. Άρα το ε, επιχείρημα της αναλογικότητας ε, μας βρίσκει αντίθετους και για αυτές τις περιόδους μεταβατικές. Εμείς προτείνουμε να προσθεθεί μια μεταβατική σε δύο ετών, ώστε να βρεθούν εναλλακτικέ για αυτή τη σημαντική ομάδα συμπολιτών μας. Ταυτόχρονα, όσο αναζητώνται αυτέ οι λύσει, να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να καταναλώνουν αυτά τα προϊόντα. Και έτσι, μετά από δύο χρόνια, η ΜΜΕ και ο κλάδος θα έχει αναπτύξει άλλε εναλλακτικέ, άλλα εναλλακτικά προϊόντα. Γι' αυτό και είμαστε αντίθετοι με την απόφαση αυτή. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Έτσι ε, ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Αύριο ψηφίζουμε. Νομίζω ότι ακούσαμε όλοι τα επιχειρήματα και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο που είναι μία αντίρρηση για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός συστήματος εχνηλασιμότητας για προϊόντα καπνού και επίσης τεχνικά πρότυπα για τα ε, χαρακτηριστικά ασφαλείας ε, που χρησιμοποιούνται για προϊόντα καπνού. Πρόκειται για μια αντίρρηση. Έχουμε πρόταση ψηφίσματος, ε, δύο ψηφίσματα συγκεκριμένα για αυτά τα θέματα. Ο κ. Πεντιτσίνη είναι ο συντάκτης αλλά έχουμε την εξή περίεργη κατάσταση. Δεν έχουμε εδώ τον ε, εισηγητή να μας παρουσιάσει τις δύο αντιρρήσεις αυτές. Άρα είτε το συζητάμε απουσία του, είτε δεν το συζητάμε το θέμα. Δεν ξέρω, θέλει κάποιος να πάρει το λόγο για την παρουσίαση της ε, αντίρρησης. Νομίζω δεν υπάρχει κανένας εδώ. Ο κύριος Φλόρενς, ο κύριος Παρνιώ και η κυρία Ζώ. Άρα μπορούμε να συνομίσουμε μεταξύ μας, απουσία του εισηγητού. Ο κύριος Φλόρεντς έχει το λόγο. Ναι. Θα ήθελα να δώσω το προβάδισμα βέβαια στον εισηγητή, αλλά αφού δεν είναι εδώ δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Πολύ σωστά είπατε ότι πραγματικά είναι κάπως περίεργο, ε, περίεργη κατάσταση. Αν διαβάσετε τα δύο αυτά έγραφα το θέμα είναι το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το καθήκον ε, να εξασφαλίσει την εχνηλασιμότητα των ε, προϊόντων καπνού, να τη διαχειρίζεται ουσιαστικά. Και έγινε μία πρόταση. Ε, και πρόσφατα τροποποιήθηκε αυτή η πρόταση και σε αυτή την πρόταση για αυτή την πρόταση κατέθεσε αντίρρηση ο κύριος Πεντιτσίν. Θα σας πω εγώ περί τίνος πρόκειται στο μέλλον οι εταιρείε που να παρακολουθούν, να πρέπει να εγγυώνται την ίχνη λασιμότητα, πρέπει να είναι ως το δυνατόν ανεξάρτητες. Δηλαδή, αν μια εταιρεία μια μεγάλη εταιρεία στο Λονδίνο, για παράδειγμα, έχει ε, με, το, με την IBM ε, σχέση εργασιακή για τη διαχείριση της μάρτης κτλ. Μια τέτοια εταιρεία δεν μπορεί ε, να αναλάβει τη σύμβαση γλασιμότητας για τη Φίλιπ μόρισε δεν ξέρω εγώ για κάποια άλλη εταιρεία. Αυτή είναι η πρόταση της Κομισιόν, δηλαδή ε, αν πάνω από 10% ε, του ετήσιου τζίρου ή παροχή υπηρεσιών μια εταιρεία είναι για μια εταιρεία παραγωγή σιγάρων ή άλλων πρωτοκομμάτων, δεν θα μπορεί να λάβει την χλασιμότητα. Οι συνάδελφοι από το EFTD τώρα τι μας λένε ότι μια τέτοια εταιρεία θα πρέπει να έχει καμία, να μην έχει καμία επαφή με τέτοιες εταιρείες, 0%. Δηλαδή οποιαδήποτε εταιρεία ε, δεν θα είναι στη θέση να αναλάβει καθήκοντα τεχνολασιμότητας. Αυτό είναι το θέμα. Αν θέλουμε να έχουμε μια σοβαρή εταιρεία, γιατί περί αυτού πρόκειται. Το μηδέν επαφή ούτε καν να δίνει ε, χαρτί για εκτύπωση από υπολογιστές. Ε, είναι λίγο υπερβολικό αυτό πιστεύω και ο στόχος είναι τελικά να καθίσταται ανέφικτο το όλο εγχείρημα. Και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα τον ανταγωνισμό. Θα υπάρξει μεγάλη ε, επίπτωση κατά του ανταγωνισμού. Μια εταιρεία μπορεί να έχει ε, κάνει κάποια ανακάψη. Δεν θα μπορεί να προχωρήσει αν έχει ε, αυτό το πρόβλημα με τη επαφή εντό εισαγωγικών με τις καπνοβιομηχανίες. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι δεν είναι ε, σωστό αυτό. Στην ε, Ιταλία παραδείγματος χάρη ξέρουμε ότι είναι τελείως διαφορετικοί λόγοι οι οποίοι έχουν κάνει τον εισηγητή να προωθήσει αυτή την αντίρρηση και όχι οι λόγοι οι οποίοι αναφέρονται σε αυτά τα έγγραφα. Γι' αυτό και ζητώ να μην γίνει δεκτή αυτή η αντίρρηση. Κύριε Σπαρνιό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι πραγματικά ε, εκτίμησα όλος ιδιαίτερο την παρέμβαση του κύριου Φλόρεντς. Μου φαίνεται πραγματικά ότι ήταν ε, πάρα πολύ σωστή ε, εγώ προεδρεύω ενός, ε, μιας άτυπης ομάδας εδώ και κάποια χρόνια ε, σε σχέση με τον κρατικό παρεμβατισμό στα προϊόντα καπνού. Εδώ και μερικά χρόνια είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχουμε κερδίσει κάποιες μάχες τον τελευταίο έτος γιατί καταφέραμε να τα καταφέρουμε ώστε να πει όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη χρηματοδότηση για την ίχνη λασιμότητα μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με το πρόσχημα της καταπολέμησης των ε, του καπνίσματος. Ε, λοιπόν, νομίζω ότι παράλληλα, ε, έχω, νομίζω ότι παράλληλα καθυστερεί η λειτουργία του συστήματος ηχνηλασιμότητας ε, και ε, υπάρχει ένα πρόβλημα συντονισμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ ενός συστήματος ανεξάρτητου ιχνηλασιμότητας, ανεξάρτητου από την ε, καπνοβιομηχανία και μάλιστα έδωσε και το νομοθετικό πλαίσιο που πρέπει να υπάρχει για να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως διατήρησε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής παρά το περίπλοκο της κατάστασης και των πιέσεων των ομάδων ε, συμφερόντων. Και νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να επικροτήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, δεν ήθελε να ε, παρέμβει στην όλη αυτή τη διαδικασία. Στην όλη αυτή τη διαδικασία. Είχε, είχαμε πολλές δυνατότητες στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου να εκφράσουμε την άποψή μας. Είχαμε κοινέ συνεδριάσεις με την Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών ε, και ε, της δικής μας Επιτροπής τον Ιούνιο του 2017. Πολλές διασκέψεις στο Κοινοβούλιο από κοινού οργανωμένες με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που μας έδωσαν τη δυνατότητα να εξηγήσουμε ε, πώς θα μπορούσε το σύστημα αυτό να είναι απολύτως ανεξάρτητο. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, που συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό στον αγώνα ε, ζήτησαν να υποστηρίξουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, γιατί κατά τη γνώμη τους το να υπάρχουν τόσες πολλές αντιρρήσεις ε, τελικά ε, το αποτέλεσμα θα ήταν να επιτύχουμε αυτό που θέλει η καπνοβιομηχανία δηλαδή να καθυστερήσει η εφαρμογή του συστήματος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ζόμερ. Πράγματι δεν είναι ε, άνετο ε, να συζητάμε ε, την αντίρρηση που έχει υποβάλει ο συνάδελφος που δεν είναι παρόν. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν ζητήματα στο σύστημα ιχνηλασιμότητας. Αλλά όχι αυτό που εννοεί ο κύριος Πεντιτσίνη. Το πρόβλημα που εγώ έχω καταλάβει ότι υπάρχει είναι ότι οι παρασκευαστές ε, τσιγάρων και που είναι και οι μικροί ε, παρασκευαστές ε, έχουν προβλήματα. Μιλάμε πολλές φορές για οικογενικές επιχειρήσεις με 10 το πολύ εργαζομένους. Μιλάμε για παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση, παράγει τσιγάρα ή πουρα. Και αυτές οι απαιτήσει για την χρηλασιμότητα θα ήταν τόσο υψηλές και θα ήταν τόσο μεγάλο το οικονομικό άχθος που δεν θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την θέσπιση και τη λειτουργία αυτού του συστήματο εχνηλασιμότητα. Δεν θα μπορούσαν από οικονομική πλευρά να το αντέξουν αυτό. Θα είχε για αυτού πολύ μεγάλη οικονομική επίπτωση. Θα έπρεπε να έχουν τα σκάνερ, του εκτυπωτέ, όλον αυτό τον εξοπλισμό και αυτέ τι συσκευέ κατά τη παραβίαση anti-tampering devices ε, θα πρέπει επίσης να προσλάβουν νέο προσωπικό και όλα αυτά κάπως να τα αποθηκεύουν τα δεδομένα αυτά και υπάρχει και ένα τεχνικό πρόβλημα για τους ε, παραγωγούς τσιγάρων ότι χρειάζεται ε, να περάσει ένα χρόνο ρήμανση αρκετών μηνών το τσιγάρο για το καπνός πρέπει κάπως να οριμάσει, να βγάλει τα αρώματά του κτλ. Αυτό μπορεί να διαρκέσει ένα χρόνο και τι γίνεται με, την, ε, με τα πρώτα αυτά καπνού συνολικά. Ε, πώς θα πρέπει να ατηρείται η χνηλασιμότητα, το μηχάνημα κτλ, κτλ. Πού έχει παραχθεί, σε ποιο μηχάνημα, όλες αυτές οι λεπτομέρειες θα πρέπει να καταγράφονται και τελικά σε ποιον ε, έμπορο παρα... Ε, ποιος έμπορος παραλαμβάνει, σε ποιον διανέμονται αυτά τα προϊόντα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα κάνουν αλλά ε, τα τσιγάρα, επαναλαμβάνω, πρέπει να οριμάσουν για κάποιο διάστημα. Και σε χονδρική πώληση κάποιος ε, φορές ε, δεν έχουν να δώσουν πολλά ε, στοιχεία. Μπορούν να πούν απλά ότι ναι, μια φορά το χρόνο τα δίνουμε στον τάδε έμπορο. Δεν μπορούν να δώσουν δηλαδή σε αυτές τις λεπτομέρειες. Είναι από τεχνικής πλευράς ε, ανέφικτο αυτό. και πολλές φορές αυτή η παραγωγή γίνεται μέσα σε μια αποθήκη γιατί εκεί πρέπει να οριμάσει ο καπνός, να οριμάσει αυτά τα προϊόντα. Η οδηγία έχει στόχο σίγουρα τον περισμό του καπνίσματος. Ε, όσοι είμαστε εδώ χρόνια ε, μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπουμε ότι πάντα αυτός είναι ο στόχος ε, ε καταπολέμηση του καπνίσματος και όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα και ε, πραγματικά το σύστημα της συχνηλασιμότητας ε, δεν είναι ένα θέμα υγείας. Ε, έχουμε να κάνουμε με άλλα θέματα που δεν έχουν κάνουν σε καμία περίπτωση με την υγεία. Και νομίζω θα πρέπει να βρει έναν ειδικό κανόνα η Κομισιόν για τους μικρούς παραγωγούς ασκευαστές τσιγάρων και πούρων, γιατί δεν θα θέλαμε αυτές οι πολύ μικρές επιχειρήσεις να κλείσουν όλες. Και η πελατεία, καταναλωτές που καταλαβαίνουν τέτοια προϊόντα είναι πάνω από 35 ετών. Δηλαδή δεν πρόκειται για κάτι το οποίο θα βλάψει τους νέους. Η χλασιμότητα ε, δεν μπορεί να ε, εξυπηρετηθεί με αυτό τον τρόπο κατά την άποψή μας και σε καμία περίπτωση δεν ξέρει ε, η Κομισιόν. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένας ειδικός κανονισμό. Επίσης να πούμε ότι Δεν υπάρχει στον τομέα αυτό λαθρεμπόριο. Δεν υπάρχει παράνομη διακίνηση. Και η όλη ε, αυτή η διαδικασία σε αυτό το στόχο έχει την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Είναι κάτι όμως που δεν παρατηρείται σε αυτόν τον κλάδο. Γι' αυτό λοιπόν ε, παρακαλώ ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετεπιτάσεως ε, να βρει έναν κανονισμό, μια εξαίρεση που να καλύπτει τους μικρούς παραγωγούς για να μπορέσουν να διατηρήσουν τις επιχείρησεις που αλλιώς θα, θα τις κλείσουν, θα βάλουν λουκέτο εάν όπως έχει σχεδιάσει η Κομισιόν τώρα εφαρμόσει αυτή την πρόταση. Δεν μπορώ να στηρίξουμε τους πέντε αστέρες με αυτά που λένε εδώ και αυτά που προτείνουν. Εγώ νομίζω ότι η μόνη δυνατότητα είναι να μην στηρίξω ε, τον ε, κύριο Πεντιτσίνη στην αντίρρησή του. Θα πρέπει να το μελετήσουμε. Τι θέλουμε. Θέλουμε να κλείσουν μικρές οικογενικές επιχειρήσεις, γιατί αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Well, thank you very much. Εμείς σας ευχαριστούμε, λέει πρόεδρος. Κυρία Κονέτσνα. Κονέτσνα, Thank you. Uh, I want to speak on behalf of Len Boylan uh, from our group. Του λέω να σας μιλήσω. Ανοίξει η πολιτική μας ομάδα, αλλά δεν μπόρεσε να παραστεί και να σας τα πει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μα φέρνει αυτέ τι εφαρμοστικέ πράξει προ έγκριση και νομίζω ότι όλοι μα εδώ είμαστε υπέρ να υπάρχει ε, μια ιχνηλασιμότητα. Να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα το οποίο να είναι αποδοτικό για αυτά τα προϊόντα και έτσι να μην έχουμε προϊόντα παραδειγμένα το οποίο στην αγορά και έτσι να προστατεύεται η δημοσία η υγεία. Αν όμω αυτέ οι εφαρμοστικέ πράξει έχουν αυτήν την μορφή, θα πρέπει να τα τροποποιήσουμε και ναι, έτσι να έρθουν τα κενά που έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν στο κείμενο. Η καθυστέρηση τη υποβολή αρμοδίω αυτών των ε, πράξεων είναι βαρύ παράληψη από πλευρά τη Επιτροπή. Έχουμε το άρθρο 106 του κανονισμού. Το κοινοβούλιο, Η δύναμη αυτού του άρθρου, μπορεί να υποβάλει ένσταση σε τέτοιες περιπτώσεις. Αντίθετα με αυτά που βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εφαρμοστικέ πράξει δεν βρίσκονται εκτό τη εντολή μα και του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ειλικρινά λυπούμε για την καθυστέρηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την υποβολή στο Κοινοβούλιο αυτών των νομοθετικών πράξεων, διότι θέλησε να μας παρακάμψει. Πάντως, έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεχθεί αυτή την ένταση και να μην δυναμητήσει το όλο σύστημα ανείχνευσης και ιχνηλασίας. Και όλα αυτά προβλέπονται από την εφαρμοστική πράξη και θα πρέπει οι διατάξεις να είναι στεγανές, οπότε σας επισημαίνω ότι θα πρέπει ταχείως να θυμιστούν κάποια, κάποια ανεξάρτητα αντικειμενικά κριτήρια για τους υπεργολάβους και να υπάρξει ένα σύστημα αποδοτικό. Ένα σύστημα το οποίο να είναι εποφελία των Ευρωπαίων και να μην ενθαρρύνει την κερδοσκοπία από πλευρά τη βιομηχανία, τη κάπνο βιομηχανία, αλλά θα πρέπει να καλύψει τι ανησυχίε μα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να θεσπίσει ένα τέτοιο σύστημα αυτό το οποίο θέλουμε. Ένα σύστημα ανεξάρτητο από την βιομηχανία. Θα πρέπει ε, να συνέλθει η Επιτροπή σε όλα τι ε, προτεραιότητέ τη και να δούμε τι θα γίνει με αυτό το σύστημα ανείχνευσης και ίχνη λασιμότητας. Οπότε θα πρέπει να δούμε, να διαπιστώσουμε αυτή την καθυστέρηση. Είναι απαράδεκτη, δεν επιδέχεται δικαιολογία. Επομένως, είναι στις του Ευρωκοινοβουλίου να φροντίζει το συμφέρον των Ευρωπαίων. Περιμένω να ακούσω σε σχέση με αυτά την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια θα δούμε τι θα κάνουμε. Η σε ευχαριστούμε για το μήνυμα του συναδέλφου. Και εδώ λέω στον κύριο Φλόρεντς. Δεν θα αλλάξει σε καμία περίπτωση ε, ούτε κατένα εκατοστό, κατένα χιλιοστό να αλλάξει τίποτα με αυτό τον ε, κανονισμό. Εγώ δεν θέλω να διαφωνήσω ε, αυτά που είπε η κυρία ε, Ρενάτε Ζόμερ για τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το τι μπορεί να συνεπάγεται αυτή. Κάτι μου είπε, αλλά δεν το κατάλαβε κυρία Ζόμερ, τέλο πάντων. Ε, υπάρχουν προβλήματα, αλλά αν υπάρχουν προβλήματα θα πρέπει ε, να κάνουν κάποιες προτάσεις οι λομπίστες που να μπορούν να έχουν κάποια χρησιμότητα. Γιατί εδώ πραγματικά τίποτα δεν θα αλλάξει, δεν θα μετακινηθεί χιλιοστός πιθαμή ε, η κατάσταση, δεν θα αλλάξει. Πραγματικά να κάνουμε αυτές τις προτάσεις, αλλά να είναι σωστές, γιατί αυτό πραγματικά εδώ είναι τελείως αβάσιμο, ό,τι λέγεται. Great. Now. Anyone else? Τέλεια. Κάνα άλλος θέλει το λόγο, όχι. Ο κύριος Μπερκόφσκι από την Κομισιόν. Thank you. First of all, Η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για τη συνεχή υποστήριξη ε, σε σχέση με το μηχανισμό εχνηλασιμότητας των καπνών. Ξεκινήσαμε με την αναθεώρηση της οδηγίας ε, για τα ε, καπνά μέχρι τώρα και τώρα προσπαθούμε να φτάσουμε στο τελευταίο σημείο του νέου, στο τελευταίο στοιχείο του νέου συστήματος, την εχνηλασιμότητα και την ασφάλεια των προϊόντων. Το προτινόμενα συστήματα ήταν αντικείμενο πολλών μελετών, συζητήθηκαν ε, διεξοδικά με τα κράτη-μέλη, πέρασαν διαδικασία διαβουλευσέων, μεταξύ των οποίων και δημόσιες διαβουλεύσεις, εργαστήρια, ανταλλαγή απόψεων, ε, οργανωμένων από αυτήν την Επιτροπή. Η διαδικασία ήταν χρονοβόρα, αλλά ήταν και απαραίτητη για να φτάσουμε σε ένα τελικό προϊόν υψηλής ποιότητας που θεωρούμε ότι βρίσκει τη σωστή ισορροπία. Προτείνει ε, πλήρη έλεγχος προς την ε, ίχνη λασιμότητα ανταπεξέρχεται στις, στα, σοβα, στα αυστηρά και, στις αυστηρές και τεχνικές προδιαγραφές ε, του πρωτοκόλου EPD, όπως επίσης και στις απαιτήσει των συνομοθετών, χωρίς να δημιουργεί επιπλέον άχρηστο βάρος, δείχνει όμως κάποια ευελιξία στις, στους μικρούς και μεσαίους φορείς εκμετάλλευσης. Πρέπει όμως να δώσουμε και κάποια ανεξαρτησία στο μηχανισμό από την καπνοβιομηχανία και πιστεύουμε ότι η πρότασή μας είναι πάρα πολύ ισχυρή ως προς αυτή την κατεύθυνση. Η ανεξαρτησία τίθεται στο επίκεντρο του, του σχεδιασμού συστήματος. Ε, υπάρχει ένα σύστημα ε, υποβολής εκθέσεων και δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να δώσουν πλήρη ορατότητα της κινητικότητας των προϊόντων και δείχνει πως ε, ε, η ανεξαρτησία των φορέων που είναι υπεύθυνοι για αυτή την ανεξαρτησία ε, ελέγχονται με έναν εφικτό και αναλογικό τρόπο. Καταρχάς, ο μηχανισμός πρέπει να τύχει μια προσέγγιση πραγματικά συστημική και αυτό νομίζω ότι το κάναμε με την πρότασή μα. Επίση πρέπει να αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι η διαδικασία μας έφτασε σε ένα σημείο ε, κατά το οποίο, αν θέλουμε να επιτύχουμε το χρονοδιάγραμμα των συνομοθετών, πρέπει να ε, προχωρήσουμε, ε, να πάει ο μηχανισμό σε ένα νέο στάδιο. Θα είναι δύσκολο, αλλά νομίζουμε ότι είναι εφικτό. Επειδή τα κράτη θέλουν 12 μήνες για ε, τα για τα, για τα στοιχεία αναγνώρισης των ε, ε χρηστών. Υπάρχει ένας κινδυνός ε, να μην ολοκληρωθεί ο, ο μηχανισμός και να πάμε πάλι πίσω στην αρχή της διαδικασίας, δηλαδή η πραγματική εχνηλασιμότητα των προϊόντων καπνού θα είναι απλώς μία προοπτική και όχι μία πραγματικότητα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Ναι, κυρία Ζόμερελα, πάρα πολύ σύντομα, γιατί δεν θέλω να ξαναρχίσει τώρα η συζήτηση. Όχι, έχω ένα ερώτημα προς τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Πώς θα εμποδίσετε τα πολύ μικρά, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής ε, τσιγάρων και πούρων ε, με την ε, υποχρεωτική επιβολή του συστήματος συχνασματός. Πώς θα την αποφύγετε. Έχετε αντιληφθεί την κατάσταση, έχετε μία ιδέα στο μυαλό σας, έχετε επαφές. Πώς θα προχωρήσετε κύριε Μπερκόφσκι. Επιτρέψτε μου να απαντήσω στην ερώτηση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εδώ κάποια τεχνικά θεματάκια πρώτα-πρώτα. Αποφάσισαν οι συνομοθέτες ότι το σύστημα θα εφαρμόζεται και σε άλλα καπνικά προϊόντα. Οπότε μιλούμε τώρα για την 25η του 24. Δεύτερον, υπάρχει μία σειρά μέτρων που θεσπίζουν τη δυνάμει του εν λόγω κανονισμού. Και έτσι διευκολύνεται το έργο των μικροπαραγωγών, ας πούμε τα χειροποίητα προϊόντα, εξαιρούνται και έχουμε διάφορες ρυθμίσεις όσον αφορά την υποβολή της κοινοποίησης και αυτό το 24 ώρο για τους μικροπαραγωγούς. Κανείς εμπορευόμενος παραγωγός δεν θα πρέπει να ξέρει πότε θα απολυθεί το προϊόν την ώρα της παραγωγής ή ε, φάσεις στην παραγωγή. Αυτό αφορά την έκδοση του τιμολογίου. Θα πρέπει βέβαια να ξέρουν όλοι όσον αφορά την πώληση και αγορά τι συντελεστής ΦΠΑ προβλέπεται. Τι να σας πω, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας πω περισσότερο, αλλά αν θέλετε να σας δώσω το υπόλοιπο στοιχεία. Ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Και ολοκληρώνουμε σε σχέση με αυτό το σημείο. Αύριο θα ψηφίσουμε για τη σχετική πρόταση ένστασης. Και η τελευταία σημερινή ένσταση που θα συζητήσουμε σήμερα αφορά την γλυφοσάτη. Με το σχέδιο εφαρμοστικής πράξης για να ανανεώσει την ε, νομοθεσία τη σχετική με την έγκριση της ενεργής ουσίας. Και πάλι η κυρία Κονέζα. Αν θέλεις μπορείς να μας κάνεις τη σχετική ενημερωτική εισήγηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ανέλαβα αυτή την ε, ένσταση εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας, της ε, αριστεράς. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί το θέμα το γνωρίζουμε καλά και άλλωστε έχουμε πανυποβάλει επανειλημμένα αυτήν την ένσταση είπαμε να μην ανανεωθεί η έγκριση για την ενεργή ουσία. Επί τη βάση της ε, πρωτοβουλίας. Θα συζητήσουμε την εβδομάδα. Θέλουμε ότι η Κομισιόν και τα κρατημέλη να έχουν κάποια ενδιάμεσα προσωρινά μέτρα, ούτω ώστε να εξεραθεί αυτή η ενεργή ουσία σε σχέση με την υπόλοιπη ρύθμιση που εγκρίθηκε στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη ότι η της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προβλέπει κάποια προσωρινά ενδιάμεσα μέτρα σε σχέση με τα τεχνικά στοιχεία. Γιατί αλλιώς θα έχουμε αβεβαιότητα, δεν θα έχουμε ασφαλή δικαίου. Και τη δίνω η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Και τότε σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε υπέρβαση αρμοδοτήτων της Επιτροπής σήμερα με τον κανονισμό, ε, τέλος πάντων είναι γνωστό τι έγινε σήμερα το απόγευμα και είχαμε 18 κρατημένοι υπέρ, 9 που δεν ε, ψήφισαν την έγκριση αυτής της ε, ανανέωσης ε, της έγκρισης κράτησε αυτή η διαδικασία μια μισή ώρα γιατί εμείς είχαμε υποβάλει τις επιφυλάξεις μας τότε που εγκρίναμε το σχετικό κείμενο στην Ολομέλεια. Οπότε συνάδελφοι λυπάμαι με αυτό που έγινε σήμερα το απόγευμα. Καταλήγουμε στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη τη γνώμη μας και τη δουλειά μας. Εμείς ήμασταν απόλυτοι. Θέλαμε να υπάρχει σταδιακή κατάργηση ε, όσον αφορά τη χρήση της γλυφοσάτης. Υπάρχει κίνδυνο στους χώρους που παίζουν τα παιδιά. Τέλος πάντων, από το 2009 έχουμε γίνει μάρτυρες ε, χρήση της γλυφοσάτης που θέτει κινδύνο την υγεία των συμπολιτών μας, των παιδιών μας. Οπότε αυτό το οποίο έκανε σήμερα η Κομισιόν και το Συμβούλιο ε, ε, οδηγεί στο να καταργηθεί η έγκριση σε πέντε χρόνια. Κάνει στροφή όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να λάβει υπόψη τις δικές μας επιφυλάξεις. Εννέα κράτη-μέλη ήταν κατά της απόφασης. Δεν το λέω αυτό υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα δεν ενδιαφέρεται για τη γνώμη μας η Επιτροπή. Αυτά τα εννέα κρατημέλη και, και αυτά έχουν πολίτες που ψήφισαν για την πρωτοβουλία. Τι θα γίνει σε πέντε χρόνια, μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θα γίνει όταν απαγορευτεί η χρήση της ουσίας σε δημόσιο χώρο. Πώς θα υλοποιηθεί αυτή η βαθμία κατάργηση, αυτό δηλαδή που συμφωνήσαμε στο Στρασβούργο. Αυτό το θέμα και σήμερα τον κόσμο. Εμείς δεν υιοθετούμε τοποθετήσεις λαϊκιστικές. Δεν ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σιωπά, δεν θέλει να τοποθετηθεί. Κυρία Γιούσο, έχετε το λόγο, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Στελαέ, να σας τα πω. Άλλωστε συμφωνούμε. Έχουμε ενώπιόν μας άλλη μία ένταση όσον αφορά την ουσία γλυφοσάτη. Δουλέψαμε σκληρά, σοβαρά, ρεαλιστικά, καλύψαμε όλες τις απόψεις και νομίζω το, το μήνυμα που στα κράτη-μέλη ήταν πολύ ισορροπημένο. Τώρα όσον αφορά τον τύπο της υπόθεσης θα πρέπει αυτό να πάει στην Επιτροπή Προσφυγών όπου τα κράτη-μέλη αποφάσισαν για αυτή την πενταετία έλαβε υπόψη την άποψή μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ε, τα, είπαμε κατά την τελευταία μας πρόταση και αυτό το οποίο τώρα θέλουμε είναι να μείνει ανοιχτό το θέμα γιατί πολύ ενδιαφέρονται γι' αυτό. Νομικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει τι θέλει. Κατάργηση ή ανανέωση. Νομικά δεν στέκει αυτή η βαθμία κατάργηση. και και το θέμα των προϊόντων που περιέχουν αυτή την ουσία, το επί της ουσίας. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει, αν θέλουν να συνεχίσουν, να δουν τι εναλλακτικέ υπάρχουν για αυτό το προϊόν. Τι μπορούν να χρησιμοποιήσουν δηλαδή οι επαγγελματίε. Τι μπορούν να κάνουν για να έχουν συγκρισιμότητα στην ποιότητα κλπ. Αλλιώ θα έχουμε άνοδο των τιμών, έχουμε επίση ε, έκθεση των παραγωγών μας στην, στον θέμα του ανταγωνισμού της παγκόσμιας αγοράς. Πάντως έχουμε τα σχετικά προϊόντα, έχουμε επίσης τους σιδηροδρόμους. Εκεί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιών, γιατί η τροχή των τρένων πρόκειται να δημιουργήσουν σπίθες και πρόκειται να έχουμε φωτιές και πυρκαγιές από όλα αυτά τα χόρτα τα ζυζάνια που φυτρώνουν γύρω-γύρω στις γραμμές. Οπότε, τέλος πάντων, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουν οι αρμόδιες αρχές και θα πρέπει το σύστημα να τροποποιηθεί, να βελτιωθεί, ε, αλλά να μην έχουμε μια κρίση εμπιστοσύνης και να μην έχουμε SAE, τις επιφυλάξεις και τις αμφιβολίες. Σας υπενθυμίζω ότι θα πρέπει τα κρατημένα να λάβουν τις ευθύνες τους. Αυτοί που έλαβαν την απόφαση. Mm. Νομίζω ότι έτσι έγινε. Οπότε κακώς άργησαν τόσο πολύ. Και θεωρώ ότι ήδη το συζητήσαμε αρκετά το θέμα. Και ακούσαμε πάρα πολλές αναλήθειες και χαζομάρες και πολλές κατηγορίες που δεν στέκουν. Ευχαριστούμε. Πότσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν ήθελα να πάρω το λόγο, αλλά θα το κάνω. Και πρέπει να διαμαρτυρηθώ. Ενάντια σε αυτήν την ερμηνεία ε, της κυρίας Δελαέ. Γιατί μπορώ να διαβάσω από το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του Οκτωβρίου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει τη σταδιακή κατάργηση ε, του της γλυφοσάτης και να μην υπάρχει καμία άδεια για τη χρήση της γλυφοσάτης μετά από μετά το 2020. Ε, το είχαμε ζητήσει αυτό, είχαμε ζητήσει μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ πάρα πολύ να το θυμηθείτε αυτό. Μην ε, παρερμηνεύετε αυτό το οποίο ενέκρινε ε, μια μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα συνεχίσω στα τσεχικά. Λοιπόν, τίποτε δεν έχω να προσθέσω. Ε, σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Κονέτσνα, εκτός από ένα σημείο. Εμείς σκεφτήκαμε να υποστηρίξουμε το ψήφισμα, γιατί το ψήφισμα του Οκτωβρίου, τεχνικός και νομοθετικός, ε, είναι πιο σωστό. Συμπεριλαμβάνει περισσότερα στοιχεία και περισσότερα επιχειρήματα, τα οποία είναι πιο σχετικά με το θέμα. Για να μην λοιπόν αποδυναμώσουμε το ψήφισμα το οποίο ε, ψηφίστηκε, υπερψηφίστηκε από 355 συναδέλφους, θα ήθελα να πω ότι θα είμαι πολύ ανοιχτός ε, ως προς αυτό και πολύ ειλικρινής. Τώρα, τι να σας πω, να αντικαταστήσουμε ένα τόσο ισχυρό ψήφισμα από ένα αποδυναμωμένο ε, ε, ε, ψήφισμα με λιγότερο έντονη διατύπωση δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Πραγματικά το λέω αυτό σε σχέση με την ερμηνεία των συναδέλφων του ΕΛΚ πώς τολμάτε πραγματικά να κάνετε τέτοια ερμηνεία ενός κειμένου το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό. Το έχω πει τόσες φορές και στα κοινωνικά μέσα και θα το ξανακάνω. Θα τα πω και στον τύπο. Λόγω του τι κάνει η κυρία Ντελαέ, ε, λόγω αυτών που κάνει η κυρία Ντελαέ, θα υποστηρίξουμε το ψηφισμά αύριο, παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε σκοπό να το κάνουμε αρχικά. Πρόεδρος. Κυρία Χάζενκαμπ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να χειροκροτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκανε τα πάντα τα κατάφερε. Έχουμε μια πλειοψηφία κρατών μελών ε, που τελικά υπέκυψε στην ε, πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Μονσάντο και αυτή η ουσία θα παραμείνει ακόμη πέντε χρόνια παρά το γεγονός ότι καταστρέφει το περιβάλλον και κυρίως είναι καρκινογόνος αυτή η ουσία. Δεν υπάρχει μάλιστα και κανένα περιορισμό χρήση τη παρά το γεγονό ότι ήταν ένα από του όρου του βασικού που είχε θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όσον αφορά τη σταδιακή κατάργηση που ζήτησε το Κοινοβούλιο, δεν υπάρχει στην πρόταση. Δεν αναφερόμαστε καθόλου στο γεγονό ότι είναι και η τελευταία άδεια χρήση αυτή τη ουσία. Είναι ένα δηλητήριο αυτή η ουσία, ένα από τα μεγαλύτερα δηλητήρια στον κόσμο ε, και για τον άνθρωπο και για τα ζώα και για το περιβάλλον. Και πολλοί πολίτες χρησιμοποιούν αυτήν την ουσία, την καταναλώνουν χωρίς το ξέρουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέτει σε κίνδυνο 500 εκατομμύρια πολίτες και τα ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρία εκατομμύρια πολίτες ε, είχαν ε, με βάση την ε, διαδικασία των πολιτών ζητήσει την κατάργησή της και εσείς το πετάξατε αυτό στα σκουπίδια. Πραγματικά ε, νομίζω ότι αυτό που κάνετε θάβει εντελώς κάθε προσπάθειά μας για κατάργηση αυτής της ουσίας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιούλκερ. Yeah. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σε σχέση με το σχέδιο ψηφίσματος και την έκκλησή του που είναι η κατάργηση της κλειφωσάτης άμεσα και να υπάρξουν μεταβατικά μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση της συγκεκριμένη ουσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να επανεισημάνω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι ότι δεν υπάρχουν ε, επιστημονικοί λόγοι που να υποστηρίζουν την κατάργηση της ουσίας αυτής στον κανονισμό για τα ε, προϊόντα φυτοπροστασίας είναι κάτι το οποίο έχει ελεγχθεί από την ΕΦΣΑ, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα ήταν αυτό ότι δεν δικαιολογείται το να ταξινομηθεί αυτή η ένωση ως καρκινογόνος. Ε, σε άλλες χώρες, στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, ε, και ε, στην ε, ομάδα για τα κατάλοιπα εντομοκτώνων του ΦΑΟ κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα. Και ο ΠΟΕ είναι ο μόνος οργανισμός στον οποίο μπορούμε να επαφιέμεθα για την ταξινόμηση της ουσίας αυτής ως καρκινογόνου. Ε, στις 9 του 2017 ε, του Νοεμβρίου του 2017 ε, υπήρξε δημοσίευση μιας μελέτης που έγινε με την έκθεση πολλών ε, εργαζομένων σε αυτή την έκθεση και το αποτέλεσμα ήταν ότι όταν χρησιμοποιείται η ουσία αυτή σε σωστή, με σωστές γεωργικές πλακτικές δεν ε, δημιουργεί κίνδυνο ε, στο περιβάλλον και στον ανθρώπινο οργανισμό. Αντιθέτως, όπως έχει υποθεί πάρα πολλές φορές στο Κοινοβούλιο και δεδομένων όλων των πληροφοριών που υπάρχουν για την γλυφοσάτη, δεν μπορούμε να θέσουμε να αμφιβόλο την επιστημονική αξιολόγηση για την ουσία αυτή, ε, η οποία έχει λάβει χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα την σταδιακή κατάργηση, εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι στο πλαίσιο του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει αυτή τη στιγμή, αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν δεν, εγκρίνεται, δεν ανανεώνεται η έγκριση, ε, η αποδοχή της ουσίας και όπως είπα για την ώρα δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία και επιστημονικοί λόγοι για να μην ανανεώσουμε την έγκριση της ουσίας αυτή. Ε, και συνεπώς ε, η ε, σταδιακή κατάργηση δεν είναι δυνατή. Βάσει της επιστημονικής αξιολόγησης και, και λαμβανομένων υπόψη άλλων ε, ε, στοιχείων όπως το ψήφισμα του Κοινοβουλίου τη 24 η Οκτωβρίου του 2017 ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανέωσε την χρήση τη ουσία αυτή για πέντε χρόνια. Αυτό είναι μια, ένα σύνδεσχρονο χρονοδιάγραμμα στις 9 Οκτωβρίου ε, το ε, ψηφίσαμε αυτό. Τα κράτη-μέλη ανέφεραν ότι θα είχαν ε, τότε εγκρίνει την ανανέωση της χρήσης ουσίας για περίοδο πάνω από 5 χρόνια. Δεδομένων όμως των νομικών υποχρεώσεων και το γεγονός ότι πληρούνται τα τα, οι προϋποθέσεις για την έγκριση της γλυφοσάτης βάσει του κανονισμού φυτοπροστασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ε, την πρότασή της στην Επιτροπή Προσφυγών ε, σήμερα το απόγευμα. Ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστηρίχθηκε από ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Again, on this objection we voted. ευχαριστώ πολύ. Θα ψηφίσουμε αύριο την αντίρρηση αυτή και εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα τις εργασίες μας. Θα σας δω αύριο το πρωί. Εννέα. Εννέα ακριβώς Καλό βράδυ, ευχαριστώ.